va, on fait la tournée nationale. Witam Państwa bardzo serdecznie. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινάμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Ας ερωτήσουμε από σεμινάριο. Ξεκινάμε από ένα σεμινάριο μία παρουσίαση δηλαδή, μίας μελέτης. Γι' αυτό και καθυστέρησα κάπως να ξεκινήσω τη συνεδρίαση, περιμένοντας στο μεταξύ να έρθουν και περισσότεροι ευρωβουλευτές. Θα ακούσουμε την παρουσίαση της μελέτης με τίτλο «Συγκριτική ανάλυση των μέσων διαχείρισης κινδύνου από το Γεωργικό Νομοσχέδιο των ΗΠΑ το 2014 και της κοινή γεωργικής πολιτικής για την περίοδο 2014-2020. Οπότε έχουμε ήδη εδώ και κάποια χρόνια εμπειρία. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποια στοιχεία όπως ε, το επίπεδο των εισοδημάτων με την εφαρμογή διαφορετικών μηχανισμών ανάλογα με τους ε, επιμέρους κλάδους της γεωργίας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη όλο το ιστορικό της, της γεωργικής πολιτικής, ε, διαφορετικές, διαφορετικά οράματα και προσεγγίσεις της ε, γεωργικής πολιτικής και στις Ηνωμένε Πολιτείε αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της μελέτης είναι μια συγκριτική ανάλυση των διαφόρων μηχανισμών και εργαλείων ε, διαχείρισης του κινδύνου που ισχύουν στις Ηνωμένε Πολιτείε, δυνάμει του Γεωργικού Νομοσχεδίου του 2014 και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και με βάση αυτή την συγκριτική ανάλυση θα αντιλήσουμε συμπεράσματα προκειμένου να προτείνουμε κατάλληλες για την Ευρωπαϊκή Ένωση λύσεις για την κοινή γεωρική πολιτική ιδιαίτερα για το ευαίσθητο θέμα της διαχείρισης των κινδύνων και την εξασφάλιση του γεωργικού εισοδήματος. Αναμένεται πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολουθεί μάλιστα την πρωινή ενδιαφέρουσα συζήτηση για το TTIP. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ζαν Κορδιέ που θα μας παρουσιάσει εκ μέρους του Γαλλικού Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών τη μελέτη αυτή. Έχει πλούσια πείρα ο εμπειρογνώμονας μας, ο κύριος Ζαν Κορδιέ. Είναι και μέλος του Agro Campus. Θα του δώσω το λόγο και χαιρόμαστε ιδιαίτερος για την ευκαιρία που θα έχουμε να ακούσουμε την ενδιαφέρουσα παρουσίαση αυτής της μελέτης από τον κύριο Κορδιέ. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για την ε, φιλοξενία σας. Είναι μεγάλη τιμή που είμαι παρόν για να παρουσιάσω την εργασία που έκανα με βάση το έτοιμά σας. Ευχαριστώ που μου το εμπιστευθήκατε, το καθήκον αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης ε, όλους μου τους συνεργάτες που με βοήθησαν σε αυτή την εργασία. Κάναμε πολλές συζητήσεις επί συγκεκριμένων και θεωρητικών θεμάτων με διάφορους συναδέλφους ε, στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταλήξουμε σε αυτή την σύνθεση. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η σύγκριση των ε, μέσων διαχείρισης κρίσεων από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού και να δούμε πόσο αποτελεσματικές είναι οι μέθοδοι αυτές. Τώρα θα μιλήσω αγγλικά γιατί επειδή είναι στα αγγλικά τα, οι διαφάνειες αλλά όταν θα αντιμετωπίσω ερωτήσεις ευχαριστούμε που μιλάτε Μα μου είπαν οι διαφάνειες να είναι στα αγγλικά. Είναι πιο εύκολο να μιλήσω αγγλικά για να παρουσιάσω διαφάνειες, αν μου επιτρέπετε. Θα μιλήσω λοιπόν σε πέντε τμήματα. Πρώτα θα παρουσιάσω... Ε, καλά, θα μιλήσω γαλλικά. Οκ, θα μιλήσω γαλλικά. Δεν θέλω να σοκάρω κανέναν. Συγγνώμη, συγγνώμη, διακόπτει ο πρόεδρο. Μια στιγμή, μια στιγμή. Κύριε Ευρωβουλευτά, ο καλεσμένος μας ανέλαβε μία εντολή, ε, το τη μελέτη και του ζητήσαμε να υποβάλει αυτές τις διαφάνειες που είναι στα αγγλικά. Από πρακτική άποψη, καλύτερο θα ήταν ε, για όλους να μιλήσει αγγλικά. Θα ολοκληρώσουμε και πιο γρήγορα το θέμα. Δείξτε λίγο κατανόηση. Τρέφουμε απόλυτο σεβασμό προς τη γαλλική γλώσσα. Μην το εκλάβετε ως προσβολή, αλλά καλύτερα αγγλικά. Ναι, αλλά κοιτάξτε, υπάρχουν διερμηνείς οι οποίοι εργάζονται θαυμάσια που θα μπορούσαν να μεταφράσουν αλλά επειδή η Γαλλία είναι η ιδρυτική χώρα της Ένωσης, μία από τις τρεις ιδρυτικές χώρες, λέει ο μιλητής, οπότε ε, ε να τη σεβόμεθα και στις νομοθετικές αρμοδιότητες και στη φύση της. Donc je vais poursuivre en français. Λοιπόν, συνεχίζω. Γαλλιστή. Έχουμε πέντε τμήματα της παρουσίασης. Πρώτα θα επενθυμίσω τους ε, συγκεκριμένους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε και τα κύρια μέσα διαχείρισης που χρησιμοποιούμε. Θα μιλήσουμε για την ε, περίπτωση των ΗΠΑ κατόπιν, μετά την ε, περίπτωση της Ευρωπαϊκής και μετά θα κάνουμε μια σύγκριση. Και αυτό που γράφουμε τον ε, αντίθετο χαρακτήρα των ευρωπαϊκών και αμερικανικών πολιτικών. Βεβαίως η ανάλυση μας επιτρέπει να καταλήξουμε σε κάποιες συστάσεις που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Οι κίνδυνοι για τη Γεωργία είναι πολλοί. Υπάρχουν κίνδυνοι αγοράς, ε, οι διακυμάνσεις των τιμών, ε, των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη γεωργία, τους κινδύνους για υγειονομικούς λόγους, τους κλιματικούς κινδύνους και όλο και περισσότερο αυτό που αποκαλούμε εξωγενείς διακυμάνσεις αλλά και ενδογενείς διακυμάνσεις που έχει να κάνει με, το χρηματοπιστω... με τις χρηματοδοτήσεις, μάλλον τις ε, τιμές των διαφόρων προϊόντων, όπως ε, το πετρέλαιο κτλ. Αντιμετωπίζουν λοιπόν όλο και περισσότερες δυσχέρειες τεχνικές, ε, εμπορικές και άλλες. Ορισμένες όμως είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη, για παράδειγμα το χαλάζι, ο παγετός, είναι αυτόνομη κίνδυνη. Μπορεί να υπάρξει παγετός εδώ και όχι εκεί. Υπάρχουν λεγόμενοι συστημικοί κίνδυνοι, όπως η τιμή που μπορεί να θίξουν οι τιμές, που μπορεί να θίξουν όλους τους γεωργούς. Από τον, στον άλλο άξονα βλέπετε τους κινδύνους ε, από πλευράς έντασης, από τους ε, φυσιολογικούς κινδύνους μέχρι τους καταστροφικούς κινδύνους. Άρα, εφόσον έχουμε τόσους κινδύνους, έχουμε και τόσα μέσα αντιμετώπισης. Κανένα μέσο δεν μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε όλους τους κινδύνους οι αυτόνομοι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται μέσω ασφάλισης, ενώ οι συστημικοί κίνδυνοι στο παρελθόν αντιμετωπίζονταν από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ε, όπως το over the counter. Επίσης, έχουμε συστήματα μέσω συνεταιρισμών για την ε, διάχυση των κινδύνων και υπάρχουν και υγειονομικοί κλιματικοί κίνδυνοι σε διάφορες χώρες. Όλα όσα προανέφερα είναι ιδιωτικού χαρακτήρα ε, μηχανισμοί που μπορούν να επιδοτηθούν από το κράτος. Τι μπορεί να κάνει το κράτος. Είναι να υπάρχει ψηλά ένα δημόσιο δίκτυ ασφαλείας, γιατί αν υπάρξουν καταστροφές, θεομηνίες, σε όλα τα κράτη-μέλη παρεμβαίνει το δημόσιο. Και επίσης μπορεί να υπάρξουν δημοσιονομικές πολιτικές που προσπαθούν, όπως και σε άλλους τομείς, να βοηθήσουν τη γεωργία. Είναι λοιπόν πολύ συγκεκριμένα τα μέσα, συμπληρωματικά και πρέπει να είναι συντονισμένα. Αυτό θα ήταν το ιδεώδες. Ποια είναι η αμερικανική κατάσταση. Εδώ βλέπετε ένα σχήμα. Υπάρχει επικάλυψη ορισμένα μέσα μπορούν να εφαρμοστούν από κοινού. Και υπάρχει πληθώρα δυνατοτήτων. Υπάρχουν οι ασφαλίσεις, ασφάλιση επί του ύψους της σοδιάς και εδώ και πολλά χρόνια παρεμβαίνουν και τα χρηματιστήρια και στη μέση, εδώ και 20 χρόνια, έχουν ε, αρχίσει να αναπτύσσονται τα λεγόμενα υβριδικά συστήματα Και από κάτω βλέπετε στο παραλληλόγραμμο ορισμένα περίπλοκα προγράμματα, δεν θα τα σχολιάσω. Έχει τις λεπτομέρειες στο κείμενο. Και πάνω πάνω, εκεί που μιλάμε για τους καταστροφικούς κινδύνους, το Αμερικανικό Νομοσχέδιο για τη Γεωργία έχει αναπτύξει αντικυκλικά προγράμματα, διατήρησε τα προγράμματα δημόσιας αντασφάλισης και μερικές ε, πληρωμές ad hoc σε περιπτώσεις εντόνων θεομηνιών. Λοιπόν, τώρα μου λείπει ένα σχήμα κάπου εδώ. Α, να το. Ο προπολογισμό. Ο προπολογισμό προβλέπει το Farm Bill, το νομοσχέδιο για τη Γεωργία. Στο τίτλο 4, διατροφή, προβλέπει επιστηστική βοήθεια. Και εδώ είναι το σημαντικότερο τμήμα του προπολογισμού, το οποίο είναι τρομερά μεγαλύτερο από όλα τα άλλα τμήματα. Αν αφαιρέσουμε την επιστηστική βοήθεια, μένουν δύο τύποι χρηματοδότηση τη γεωργίας από το δημόσιο, κυρίως τα υβριδικά ασφαλιστικά συμβόλαια και κατόπιν τα αντικυκλικά προγράμματα και άλλα και άλλα δημόσια προγράμματα που είναι αποκλειστικά δημόσια και όχι ιδιωτικά με μια δημόσια ενίσχυση. Ο προπολογισμό λοιπόν ε, των ΗΠΑ αφορά, συγγνώμη, εμπλέκεται και στα ιδιωτικά συμβόλαια. Αυτά τα συστήματα είναι πλήρη, αλληλοσυμπληρούμενα και δυναμικά. Αυτό που μάλλον δεν υπάρχει είναι τα φορολογικά μέτρα, τα φορολογικά κίνητρα. Και όταν έθεσα το ερώτημα, γιατί δεν υπάρχει αυτή η βοήθεια, για παράδειγμα, στην προληπτική αποταμίευση. Μου είπαν ότι δεν ασχολείται με αυτό το Υπουργείο Γεωργίας, αλλά το Υπουργείο Οικονομικών, οπότε γίνεται αλλού συζήτηση. Αλλά έχω δει μελέτες που θεωρούν ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Η ανάλυση δείχνει ότι η διαχείριση κινδύνων γίνεται με δύο πυλώνες, με δύο διαφορετικούς κανονισμούς, 1305 και 1308, θα ξαναμιλήσουμε για, αυτές, για αυτούς τους κανονισμούς. Άρα ήδη υπάρχει μια διέρεσε δύο. Η ανάλυση μου είναι ότι οι τεχνικές παράμετροι του δικτύου ασφαλείας δεν είναι τεχνικές. Δεν θα έλεγα ότι ε, στρεβλώνονται, αλλά είναι συζητήσιμες, επηρεάσιμες. Και δίνω ένα παράδειγμα μέσω της ε, αντιμετώπισης του ρωσικού εμπάργου για το πώς χρησιμοποιήθηκε το αποθεματικό. Αν το βλέπει κανείς από τα έξω ως ε, πρωτοασχολούμενος με το θέμα αυτό, του φαίνεται αρκετά καταστροφική η διαχείριση. Λοιπόν. Υπάρχουν τρία άρθρα που αναφέρονται στο νένα πυλώνα για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις ε, ασφαλίσεις αν υπάρξουν σημαντικές απώλειες πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν αμοιβαία κεφάλαια για τους κινδύνους σοβιάς και κατόπιν έγινε μια αντιγραφή του άρθρου 38 στο άρθρο 39 με κάποιες τροποποιήσεις και στο άρθρο αυτό λέγεται ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν δημόσια, συγγνώμη, αμοιβαία κεφάλαια για να βοηθήσουν την γεωργία. Από το 2005 έχει μελετηθεί κατά πολύ αυτή η λύση αλλά δεν έχει εφαρμοστεί. Γι' αυτό λέω ότι είναι θεωρητική αυτή η αντιμετώπιση. Είναι ένα ιδιαίτερο είδο ε, κατάσταση. Επιπλέον, η ερμηνεία των κειμένων γίνεται με πολύ αυστηρό τρόπο. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκα για κάποια αμοιβαία κεφάλαια στη Ρουμανία και συζητάμε για να ορίσουμε τι είναι απώλεια παραγωγής. Είναι απλό. Μιλάμε για απώλεια όγκου, κύκλου εργασιών, δεν ξέρουμε. Ακόμη δεν έχουμε καταλάβει. Πώς λοιπόν να εφαρμόσει κάτι όταν δεν έχεις τα στοιχειώδη. Και για διάφορους λόγους, λόγω της ποικιλία των ε, υγειονομικών και κλιματικών κινδύνων υπάρχει πολύ μεγάλη ανομοιογένεια του συστήματος. Βλέπετε εδώ μια ιμπρεσιονιστική εικόνα της ανομοιογένειας που δείχνει ότι θεωρητικά υπάρχουν ε, ορισμένα μέτρα που δεν εφαρμόζονται, ότι υπάρχει, δεν ξέρουμε πώς εφαρμόζεται και αν θέλαμε να περιγράψουμε τη γεωργία στις χώρες αυτές δεν θα μπορούσαμε. Έχουμε ιδιαίτερε περιπτώσεις ο βορράς της Ευρώπης, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία που έχουν αναπτύξει κάποια αμοιβαία ταμεία, η Ισπανία και η Αυστρία που έχουν αναπτύξει κάποια συστήματα εκτός επιδοτήσεων και η Τουρμανία που ξέρουν προσπαθεί επίσης να δημιουργήσει ένα σύστημα. Είναι λοιπόν μπαλώματα. Σύγκριση. Οι πολιτικές αυτές είναι διαφορετικές είναι στις δύο άκρες ε, της κλίμακας. Αν δείτε ε, εδώ στον πρώτο πίνακα πόσο μακροσκελή είναι τα κείμενα και στο δεύτερο το ύψος του προπολογισμού. Τα ίδια λένε οι δύο πίνακες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η γεωρική πολιτική για τη διαχείριση των κινδύνων είναι το, το πρωταρχικό, η βοήθεια στη διαχείριση κινδύνων. Κατόπιν έχουμε τα δίκτυα ασφαλείας και όπως ξέρετε έχουν καταργήσει την, ε, τις άμεσες πληρωμές, την ενίσχυση του εισοδήματο το 2014. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζει την ε, πολιτική της στις άμεσες πληρωμές, ενίσχυση του εισοδήματο, λέγοντας είναι ίσως ε, και μέσω διαχείρισης κινδύνου, πουθενά δεν έχει, δεν έχει υποθεί σαφώς, αλλά δεν είναι ασφάλιση κάτω του κινδύνου. Το μεγαλύτερο τμήμα του προπολογισμού λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ασχολείται με διαχείριση κινδύνων. Υπάρχει χρηματοδότηση των δικτύων ασφαλεία 5% και η συγκεκριμένη βοήθεια για τη διαχείριση κινδύνων είναι απόλυτα μελιτέα. Θα αυξηθεί ερώτηση. Η εντύπωσή μου είναι ότι στη σημερινή συγκυρία δεν θα αναπτυχθεί, άρα κάτι πρέπει να γίνει. Οι πίνακες είναι κάπως σχηματικοί, αλλά νομίζω ότι καταδεικνύουν την κατάσταση. Επιπλέον, στις Ηνωμένε Πολιτείες, τα μέσα διαχείρισης κινδύνων και τα δίκτυα ασφαλείας <clears throat> συνδυάζουν την δράση τους. Οι ίδιες παράμετροι ορίζουν την καταστροφή, του τι σημαίνει αποδεκτός κίνδυνος, τι μπορεί να, δηλαδή, να αναλάβει να καλύψει ο ιδιωτικό τομέα ως κίνδυνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει κανένας ορισμός. Στον πυλώνα 1 και λίγα πράγματα στον πυλώνα 2. Η κοινή, συγγνώμη, η αμερικανική γεωρική πολιτική έχει ορισμένα πλεονεκτήματα. Το κύριο είναι ότι δημιουργεί βάσεις δεδομένων. Έχει εδώ και χρόνια συλλέξει εμπειρία και βασίζονται στη γνώση. Και αυτό είναι για μένα το μέλλον. Και το αντίθετο είναι οι άμεσες πληρωμές. Όπου στην ουσία μοιραζόμαστε μια πίτσα και ο καθένας προσπαθεί να πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι. Ο στόχος της διαχείρισης των κινδύνων είναι να αυξηθεί η παραγωγή, ούτως ώστε όλοι να υποφεληθούν. Δεν είναι λοιπόν της ίδιας διάστασης συμβολή στην κοινότητα. Το αρνητικό του αμερικανικού προτύπου το έχουμε διαπιστώσει. Είναι ότι οι γεωργοί πηγαίνουν προς την κάντιλακ των ε, ασφαλίσεων. Δηλαδή η ευρύτερη κάλυψη κινδύνων με πολύ χαμηλά ασφάλιστρα λόγω της επιδότησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει. Το άρθρο 37 και 38 και τη διαχείριση των κινδύνων και το 39 για τις ε, μορφές ε, αμοιβαίας σταθεροποίησης των εισοδημάτων είναι κατά την άποψή μου καλές βάσεις. Ωστόσο, η ερμηνεία και ο τρόπος με τον οποίο βλέπω τη συμπεριφορά αυτή σημαίνει όπου ο καθένας ανοίγει την ομπρέλα του για να προστατεύεται ο ίδιος, η Επιτροπή που θέλει να είναι clean σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς εμπορίου. Τα κράτη-μέλη αφετέρου που λένε εγώ δεν θέλω να έχω προβλήματα με την Κομισιόν και έχω βιώσει αυτή την κατάσταση. Ο καθένας προσπαθεί να προστατευτεί και δεν γίνεται τίποτα. Και η η πολιτική, η ευρωπαϊκή πολιτική γεωργίας ε, κινδυνεύει να βγει σε ένα διέξοδο. Τώρα, τι μέλη γενέστε. Ξέρουμε ότι οι άμεσες πληρωμές πηγαίνουν κατευθείαν στην παραγωγή. Αυτό το λέει το οικονομικό συμφέρον. Οι, άμεσες, οι απευθείας πληρωμές λοιπόν έχουν, ε, ε, πλουτίζουν αλλά δεν περιλαμβάνουν κίνδυνο. Κατόπιν περνάει στους παράγοντες παραγωγής και η κατανομή δυσχεραίνει όταν μειώνεται το ποσό. Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα πολιτικής ωστόσο. Η γεωργική πολιτική τώρα της Ένωσης, κατά την άποψή μου, δεν έχει πραγματικό όραμα διαχείρισης κινδύνου για τους δύο πυλώνες. Δεν έχει κάποια, κάποιο όραμα. Δεν το βλέπω. Είναι δύο ξεχωριστές καταστάσεις που δεν συντονίζονται. Πώς θέλετε μεταξύ καταστροφών και απλή, απλής, διαχείριση, απλής διαχείρισης κινδύνου να υπάρχει συντονισμός. Άρα συζητούμε το θέμα από το 2005 αλλά συντονισμός δεν υπάρχει πέραν της απλής ε, επικόλυσης. Τέλος, είναι δύσκολο να διαχειριστεί κανείς έναν κίνδυνο με έναν σταθερό προϋπολογισμό. Δεν, δεν είναι δυνατό. Χωρίς να υπάρχει ευελιξία, δεν μπορούμε να μιλούμε για διαχείριση κινδύνου. Διαπιστώ, έγινε η διαπίστωση. Φτάνω τώρα στις προτάσεις, στις συστάσεις. Τέσσερις ομάδες. Πρώτον, καταρχάς να συμπληρώσουμε τα υφιστάμενα εργαλεία. Η δεύτερη ομάδα συστάσεων είναι όταν υπάρχουν λύσεις επί χάρτου πρέπει να υλοποιηθούν, δεν αρκεί να γράφουμε κάτι και μετά να λέμε κάντε ό,τι θέλετε, ε, πρέπει να γίνουν πειράματα, πιλωτικά τεστ. Η διαχείριση κινδύνου δεν έχει εκ άνω προς τα κάτω, πρέπει να ξεκινά από την ε, τοπική αλληλεγγύη που θα δημιουργήσει συστήματα με, ένα, με μια κοινή επικάλυψη που θα επιτρέπει συντονισμό και σεβασμό των αρχών λειτουργίας της Ένωσης, το fair competition κτλ. Χρειάζονται ανθρώπινοι, κατάλληλοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι που θα είναι ευέλικτοι και τέλος χρειάζεται οργάνωση. Πρώτη σύσταση, συντονισμός του, των δικτύων ασφαλείας και των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου των ιδιωτών με υποστήριξη του, της πολιτείας, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να καλυφθεί το κενό. Θα δείτε στο κείμενο αυτό, αυτό το τεράστιο κοινό μεταξύ ασφαλειών αφενός που περιορίζονται στην παραγωγή και χρηματοοικονομικών εργαλείων αφετέρου. Αυτό το κενό, το gap, πρέπει να μπορεί να καλυφθεί με το εργαλείο e IST, σταθεροποίηση εισοδημάτων, που υπάρχει όμως μόνο θεωρητικά προς το παρόν. Και πρέπει να δημιουργήσουμε εισόδημα προφύλαξης, αυτό το, που είναι μια καλή μορφή προστασίας της επερχόμενης συγκομιδής και περιλαμβάνει και ένα στοιχείο διαχείρισης κινδύνου. Δηλαδή να αποφορολογικοποιήσουμε τα αποτελέσματα, να μην φορολογούμε δηλαδή τέτοια αποτελέσματα. Αυτό έχει ένα δημοσιονομικό εθνικό ή κοινοτικό αποτέλεσμα, αλλά οι χώρε που το έκαναν θα μπορούσαν να πούν ότι η φορολογική, η δημοσιονομική υποστήριξη που κάνουμε μπορεί να θεωρηθεί ω συγχρηματοδότηση. Να υπολογιστεί δηλαδή υπομορφή συγχρηματοδότηση. Ανάπτυξη εργαλείων λοιπόν. Δεύτερη ιδέα. Να δημιουργήσουμε πιλωτικά σχέδια. Γιατί. Όπως είπα η πρωτοβουλία πρέπει να έρθει από τις επιτόπιες δράσεις. Ο μικρός γεωργός θα κληθεί, πολλοί θα σας πούν ότι πρέπει να λειτουργήσουμε με αντικυκλική προσέγγιση, θεωρητικά, σαν επικάλυψη. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Αντίθετα, το να κάνουμε τοπική αντικυκλική πολιτική, δηλαδή στη βάση των τοπικών, της τοπικής αλληλεγγύης, σημαίνει ότι κρατάμε κάτι ε, στην άκρη για τις δύσκολες στιγμές. Αν έχουμε μια μεγαλύτερη ε, θεομηνία μπορεί να φτάσουμε και στην δημόσια παρέμβαση. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει και μια τοπική κινητοποίηση. Εγώ ξέρω ομάδες και στη Γαλλία και αλλού που, έχουν αυτοί, που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο θα ήταν ενδιαφέρον να τα υποστηρίξουμε. Με τα τεστ αυτά πρέπει να μάθουμε και να δημιουργήσουμε ενδεχομένω αν χρειαστεί τι παραμέτρου που χρησιμοποιούνται στα λιμάνια, στις μεγάλε καλλιέργειε για τα αποδοκιπευτικά, για κάθε κλάδο, ε, η κατάσταση είναι διαφορετική. Δεν υπάρχει δηλαδή κοινή πρακτική. Πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχα διαφορετικά εργαλεία προσαρμοσμένα στην κατάσταση και στην τοπική πραγματικότητα. Ίσως να χρειαστεί να μειώσουμε κάποιες δεσμεύσεις που έχονται εκ των άνω για να επιτρέψουμε αυτά τα τεστ. Η τρίτη ομάδα συστάσεων. κατάλληλη ανθρώπινη και χρηματοοικονομική πόρη. Για τους ανθρώπινους ε, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. ως πανεπιστημιακός, ε, όπως όλοι οι πανεπιστημιακοί, μπορούμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία δικτύων ε, για την συνεργασία και καταμερισμό εμπειρία, στατιστικών και άλλων δεδομένων. Πρέπει δηλαδή στην ε, σοφροσύνη των ντόπιων να προσθέσουμε και λίγο τεχνογνωσία πανεπιστημίου για να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Αυτό δεν στοιχίζει πολλά, μπορεί να γίνει εύκολα, υπάρχει στην πράξη. Χρειάζονται πόροι, οικονομικοί πόροι τώρα. Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να βρεις χρήματα. Πρέπει να έχουμε ευέλικτο τρόπο μέσω των αμέσων πληρωμών ενδεχομένω. Όσο αναπτύσσονται, αργά-αργά θα αναπτύσσονται οι παράγοντες διαχείρισης κινδύνου, θα αυξάνεται η ικανότητα του αποθεματικού, επιτρέποντας μια αντασφάλιση του συστήματος διαχείρισης κινδύνων. Εγώ λέω 10% των άμεσων πληρωμών να μπουν στο αποθεματικό, αλλά αυτό είναι ένα νούμερο έτσι, μόνο και μόνο για να έχουμε μια εικόνα. Μπορεί να σας αρέσει. Τέλος, οργάνωση. Να υπάρχουν δύο πυλώνες για τη διαχείριση κινδύνου. Το να υπάρχουν μάλλον δύο πυλώνες για τη διαχείριση κινδύνου δεν στέκει. Να φέρουμε τώρα στον πυλώνα ένα τη διαχείριση κινδύνου, να δημιουργήσουμε ένα τρίτο πυλώνα, δεν ξέρω. Πάντως χρειάζεται ένας χωριστός, μια χωριστή δομή που θα κατευθύνει τη διαχείριση κινδύνου. Και γι' αυτό πρέπει να είναι ανεξάρτητος ο φορέας. Να μην πιέζεται από κινήματα, χρειάζεται να υπάρχουν τεχνικές βάσεις, ε, κανόνες που έχουν τεθεί εκ των προτέρων και εφαρμογή τους. Αυτό υπάρχει από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει το Risk Management Agency. Μια τέτοια δομή. Δεν θα πρέπει αυτός ο φορέας να είναι κάτι μελλοντικό, δηλαδή κάτι που να έχει μια προοπτική δεκαετίες, 20 ετίες, αλλά να λειτουργεί και βράχει πρόθεσμα. Να παρακολουθεί τα πιλωτικά σχέδια που θα αναδειχθούν στις διάφορες χώρες. Να παρέχει εμπειρία και τεχνογνωσία στις χώρες μην ξεχνάτε ότι η ομάδα των 20 δημιούργησε μια αντίστοιχη πλατφόρμα για τι αναπτυσσόμενε χώρε, όπου ε, γίνεται γνωστή η εμπειρία που έχει κάθε χώρα και οι βέλτιστες πρακτικές και που θα ε, διαπιστώνει κατά πόσον το κόστο διαχείριση, το management cost δηλαδή, δεν θα παίρνει τα πάνω του. Υπάρχουν τεχνικέ και μέθοδοι για την αρχιστοποίηση τη δημιουργία εργαλείων και τη λειτουργία του. Αυτά. Επίσης, Πρέπει να ελέγχουμε κατά πόσο τα εργαλεία αυτά πηγαίνουν στη σωστή κατεύθυνση, ε, λαμβάνοντας υπόψη και τα τοπικά και τα γενικά, δηλαδή την αλλαγή του κλίματος, θέματα ουσίας, ενώ μπορεί να βάλουμε και προϋποθέσεις τα εργαλεία αυτά, ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη η πρόληψη, η ανάγκη πρόληψης, η ανάγκη προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές και όλα αυτά. Εγώ το έκανα στο Μαρόκο αυτό. Αυτά Αυτές οι τέσσερις ομάδες συστάσεων είναι νέες πιστεύω και ελπίζω ότι μπορεί να σας φανούν προκλητικές σε κάποια στιγμή αλλά είναι χρήσιμες και πιστεύω ότι θα βοηθήσουν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας, είμαι έτοιμος να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Λουαζό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον εμπειρογνώμονα, τον κύριο Κορδιέ, για την παρουσίαση. Ε, δεν μπορεί κανεί να πει ότι οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται για την γεωργία του. Έχουν πολύ πιο προστατευτικά μέτρα από ό,τι εφαρμόζουμε εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί οικονομολόγοι και εμπειρογνώμονε θεωρούν ότι τα, τα μέτρα είναι και κατά του ΠΟΕ. Και μάλιστα είναι σκαδαλώδη αυτή η αφιλεγόμενη πολιτική των ΗΠΑ που συνεχίζει τι διαπραγματεύσει με, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το TTIP και ταυτόχρονα ενισχύει την προστασία των δικών τη γεωργών. Θα πρέπει να καταγγείλουμε αυτή την πολιτική. Ε, γιατί να μην αναστείλουμε και όλα τις διαπραγματεύσεις του TTIP. Επίσης, ε, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν καταφέρει να είναι ταυτόχρονα, μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση καταφέρει να είναι και, και βεβαρημένη. Νομίζω ότι κανένα δεν θα ήθελε μια τέτοια πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν άλλες φιλοδοξίες από το να μας απογυμνώσουν ουσιαστικά, να μας ξεγυμνώσουν ε, αφήνοντας μας έρμεο απέναντι στους ανταγωνιστές μας που είναι και εταίροι μας. Δεν είναι αυτοκτονική αυτή η πολιτική. Θα πρέπει να, τη δεχόμαστε, να δεχόμαστε τέτοιους παραλογισμούς με το χαμόγελο και αδιαμαρτύρητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να διακόψουμε τις διαπραγματεύσεις στο TTIP. Γι' αυτό και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αν κάνει τις διαπραγματεύσεις για τη γεωργική πολιτική να το κάνει το συντομότερο δυνατό και να μην περιμένει ε, τις υπόλοιπες διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι είναι κατεπήγον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε μία αντιπροσωπεία γεωργών από τη Σλοβακία. Ε, και μάλιστα και την Υφυπουργό Γεωργίας ε, της ε, Σλοβακίας. Καλωσορίζω θερμά την Υφυπουργό και την Αντιπροσωπή από τη Σλοβακία. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή και σας εύχομαι καλή ακρόαση των, της συνεδρίασης. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σένερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις μόνο προς τον εμπειρογνώμονα για να βεβαιωθώ ότι κατάλαβα καλά. Μετά από 25 λεπτά παρουσίασης ε, έχω κάποιες απορίες. Τι μας προτείνετε, να, αφήσουμε, να βγάλουμε το 10% των άμεσων ενισχύσεων που πηγαίνουν στο Γεωργό και να το αφιερώσουμε, σε, να το δώσουμε σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις για να διαχειριστούν τον κίνδυνο, αυτό μας προτείνετε. Δεύτερον, προτείνατε να μας βοηθήσουν τα πανεπιστήμια για να αναπτύξουμε τέτοια μέσα διαχείρισης κινδύνου. Και αν ναι, πόσο θα μας τυχήσει μια τέτοια ανάθεση της διαχείρισης του κινδύνου στα πανεπιστήμια. Γιατί νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα θαυμάσιο επιτελείο υπαλλήλων και μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το τεχνικό έργο. Μήπως θέλετε να βρεθούν κονδύλια για να, για να χρηματοδοτηθούν τα πανεπιστήμια μέσω της έρευνας για τα, για τα μέσα διαχείρισης κινδύνου. Έτσι προσπαθείτε να μας ετοιμάσετε για την κανονιστική σύγκληση όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του TTIP με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστώ. Κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα η εισήγηση του ομιλητή. Ακούσαμε πολλά νέα πράγματα. Όπως και κλειμένος μας σωστά είπε ότι δύσκολο μπορεί να, καταλάβει, να φανταστεί κανείς μια κατάσταση που θα μπορέσουμε να, να συνεχίσουμε να υπάρχουμε χωρίς απευθείας άμεσες πληρωμές. Ωστόσο, τα κονδύλια η, αρχικά τα αγροκτήματα ήταν λίγα, οι, ομάδο, ομάδες παραγωγών περιορισμένες, είχαμε μικρούς ε, παίκτες στην αγορά. Άρα οι ε, άμεσες ενισχύσεις λειτουργήσαν, λειτουργούσαν. Μπορούσαν να πάρουν οι, ε, ε, επαρκές εισόδημα οι γεωργοί μας και να εξασφαλίσουν τα προστοζήν για τον, τους αυτούς και την οικογένειά τους. Σήμερα ωστόσο, αν δούμε τις διάφορες χώρες θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν διαφορετικών μεγεθών επιχειρή, αγροκτικές επιχειρήσεις στην Λιθουανία. Υπάρχουν τέσσερις, ε, τέσσερις, ε, τέσσερα εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων. Ε, στην πραγματικότητα λειτουργούν υπό μορφή καρτέλ. Πώς μπορούμε να εμποδίσουμε τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ από το να κερδοσκοπούν αφαιρώντας ε, το ποσοστό, ποσοστό εισοδήματος των γεωργών. Εμείς έχουμε τώρα το εμπάργκο της Ρωσίας. Βλέπουμε ότι οι τιμές ε, του γάλακτος έχουν αυξηθεί δραματικά. Στα, στο γιανεμπόριο ωστόσο, δεν μειώνεται η τιμή. Οι γεωργοί παίρνουν εθνική ενίσχυση, παίρνουν ευρωπαϊκή ενίσχυση, η ενίσχυση αυτή μειώνεται, διότι οι τιμές αγοράς πέφτουν και αυτές. Εν τέλει, οι γεωργοί καταφέρνουν να επιβιώσουν χωρίς να κερδίζουν ωστόσο και στον τομέα του κρέατος και στα γαλακτοκομικά. Το σύστημα άμεσων ενισχύσεων μπορεί να παρέσχει γενικά ισότιμη προστασία. Μπορούμε να πούμε ότι ένας νέος θα θέλει να ξεκινήσει αγροτικές δραστηριότητε. Ένας γεωργός μπορεί να έχει μια εικόνα πώς θα είναι σε 10-15 χρόνια η γεωργική του εκμετάλλευση. Αυτά είναι τα ερωτήματα που αντιμετωπίζουν οι ε, γεωργοί. Τώρα για τις τιμές αγοράς, αν επιτρέψουμε να, να αδράτουν τα κέρδη οι μεσάζοντες, τι θα γίνει με τα χρήματα των φορολογούμενων, θα, θα ενισχύουν τους πλούσιους, όχι αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. Εγώ συναντήθηκα πρόσφατα με την Ένωση Γαλακτοπαραγωγών της Λιθουανίας και Μάλιστα αυτές, αυτές τις μέρες γίνεται και ένα συνέδριο των παραγωγών στην Λιθουανία. Πρότειναν ένα νομοθετικό κείμενο για ρύθμιση τιμών εφόσον οι τιμές δεν είναι ε, ρυθμισμένες, οι άμεσες ενισχύσεις χάνουν τη σημασία τους. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς ε, αυτά που προτείνεται για να εξετάσει τα υπέρ και τα κατά της πρότασής σας. Θα πρέπει να σκεφτούμε ωστόσο την καλύτερη εναλλακτική λύση για μας στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νταντά. Παρακαλώ κύριε Νταντά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για την ε, παρουσίασή σας. Όταν η Επιτροπή Γεωργίας εξέτασε το θέμα της ε, ενισχύ ΚΓΠ, δημοσιεύτηκε μια έκθεση του Αμερικανικού Κογκρέσου που έδειχνε ότι για κάθε δύο δολάρια που επενδύει το Αμερικανικό κράτος οι γεωργοί λάμβαναν 0,8 μέσω της πολιτικής διαχείρισης και κάλυψης των κινδύνων. Σε τι βαθμό η νέα Αμερικανική γεωργική πολιτική τροποποιεί αυτή την κατάσταση για να βελτιώσει την απόδοση αυτών των ε, δημοσίων αμερικανικών επενδύσεων, την αύξηση δηλαδή του ποσού που λαμβάνουν οι γεωργοί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κουτενάνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ ειλικρινά τον κύριο καθηγητή για την παρουσίασή του, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια σύγκριση της κατάστασης ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες με την κατάσταση στην Ένωση. Δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε την κοινή γεωρική πολιτική που νομίζω ότι έχει αποδείξει την αξία της. Επέτρεψε την επιστηστική επάρκεια στην Ευρώπη. Μας επέτρεψε να αναπτύξουμε προϊόντα ποιότητας και δεν μπορούμε να την καταργήσουμε έτσι με μια χειρονομία. Και δεν νομίζω ότι αυτή η σύγκριση στην ουσία αποβαίνει υπέρ των ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτά που επιτύχαμε στην Ευρώπη. Και να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Ωστόσο, ωστόσο, φυσικά δεν θα παραμείνουμε στάσιμοι. Το θέμα του ασφαλιστικού είναι ουσιώδες. Πρέπει να το δούμε για την επόμενη κοινή γεωρική πολιτική. Διότι μέσω των ασφαλίσεων μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κρίσεις που έχουν προκύψει τοπικές, ε, ευρύτερες να μην ξεχνάμε ποιος ο στόχος μας να θρέφουμε τους πολίτες μας και τον πλανήτη και να έχουμε γεωργικά προϊόντα που να είναι αντάξια των προσδοκιών μας και οι γεωργοί πρέπει να μπορούν να ζήσουν από την γεωργία. Αυτή είναι η ουσία. Βεβαίω θέλουμε τρόφιμα υψηλή ποιότητα, αλλά πρέπει και οι γεωργοί να μπορούν να ζήσουν. Σωστά, αξιοπρεπώς. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Άρα το, οι το ασφαλιστικό πρέπει να το δούμε. Και σα ευχαριστώ που το θέσατε. Είπατε 10%. ε, υπήρξαν αντιδράσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το δούμε ε, πιο αναλυτικά. Ευχαριστώ κύριος Ντόφμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτό που υπόθηκε είναι πολύ ενδιαφέρον διότι όντως σε αυτή τη συγκυρία πρέπει να σκεφτούμε πώς μέσο και μακροπρόθεσμα θα προχωρήσει η κοινή γεωρική πολιτική. Είμαι από μια περιοχή στην οποία υπάρχουν πολλές ασφαλίσεις, άρα δεν συμφωνώ ότι δεν υπάρχει καθόλου ασφαλιστική κάλυψη. Και υπάρχει μεικτή χρηματοδότηση. Αλλά έχετε δίκιο. Αν θέλουμε πραγματικά να υπάρχει σταθερό εισόδημα των γεωργών, πρέπει να υπάρξει πολύ ευρύτερη χρηματοδότηση. Δηλαδή, το σημερινό σύστημα των αμέσων πληρωμών θα μπορούσε να αντικατασταθεί με ένα σύστημα ασφαλίσεων. Θα κάνουμε ή το ένα λοιπόν ή το άλλο. Αν δούμε τι έχει γίνει σε ορισμένους τομείς της γεωργίας τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα ποιες επιφάνειες ε, καλλιεργούνται, τότε θα πρέπει να δούμε εάν όντως χρειάζονταν όλοι οι παραγωγοί αυτές τις άμεσες πληρωμές. Διότι όλο και περισσότερο θα έχουμε ε, περιπτώσεις που πολλές επιχειρήσεις μπορούν να ζουν χωρίς να παράγουν. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν τομείς όπως ε, ο γαλακτοκομικός όπου είναι πολύ χαμηλό το εισόδημα σε αυτούς θα μπορούσαμε να δούμε πω κάποια στοιχεία του αμερικανικού προτύπου θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν για να απτύξουμε περαιτέρω την γεωργική μας ε, πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μαγκίνες. Και ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Θα πρέπει φυσικά να την εξετάσουμε πιο διεξοδικά, γιατί ήταν πολύ σύντομη η παρουσίαση. Από τη πιο σημαντική ε, φράση είναι στη σελίδα 53. Μιλάτε για τις διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, τις δημοσιονομικές και ότι ο δικός μας προϋπολογισμός είναι πάγιος και περιορισμένος. Κάτι που δεν ισχύει για τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν πιο ελαστικό προϋπολογισμό και αναλαμβάνω σε μεγάλο βαθμό τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της διαχείρισης κινδύνου και των μέσων και των δικτύων ασφαλείας. Θα ήθελα να μας αναπτύξετε αυτό το σημείο. Πολύ εύστοχα και τα σχόλια του κυρίου Ντόρφμαν. Και ατενίζοντας το μέλλον, διαπιστώνουμε ότι θα πρέπει στο μέλλον να λάβουμε πολύ ε, δύσκολες αποφάσεις και θέλουμε καλύτερη καθοδήγηση για το τι είναι αποτελεσματικό και τι όχι. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε οικογενειακές ε, εκμεταλλεύσεις. Μας ενδιαφέρει η υπεθρός και στηρίζουμε την ανάπτυξη της υπέθρου την αγροτική ανάπτυξη και τέτοιου είδους πληρωμές ε, και ενισχύσεις είναι σημαντικό να στηρίξουν την υπεθρό. Τώρα ε, νομίζω ότι όταν σχετίζονται οι άμεσες ενισχύσει με τη γη, ουσιαστικά κεφαλαιοποιούν το κόστος. Και δεν νομίζω να βοηθούμε τόσο πολύ έτσι τους ε, παραγωγούς, γιατί δεν στηρίζονται τόσο στην παραγωγή. Επίσης, αν λέτε το 10% των άμεσων ενισχύσεων να το αφαιρέσουμε από τους γεωργούς για να δημιουργήσουμε μια πολιτική ασφαλίσεων, δεν ξέρω, είναι ένα πολιτικό το δίλημα. Εσείς ε, πού πιστεύετε ότι βρίσκεται το μέλλον της Ευρώπης για τη Γεωργία. Είπατε ότι δεν έχουμε όραμα. Έχουμε όραμα, αλλά δεν έχουμε μέσα για να το υλοποιήσουμε. Και θέλουμε και τον κατάλληλο προϋπολογισμό για να πραγματοποιήσουμε το όραμά μας. Μπορείτε να τα αναπτύξετε και αυτά παρακαλώ στην απάντησή σας. Νομίζω ότι έλαβαν το λόγο όσοι τον είχαν ζητήσει. Οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Χανιώτη της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη και να μας κάνει κάποια σχόλια μετά την παρουσίαση και το εμπειρογνώμονα και ενδεχομένως και να απαντήσει στις ερωτήσεις. Oh, thank you, Σας ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω το λόγο στον εμπειρογνώμονά μας. για να απαντήσει ενδεχομένω και αυτός στις ερωτήσεις. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Και θα προσπαθήσω να τις ομαδοποιήσω για να απαντήσω καλύτερα. Δεν θα έλεγα ότι το μέλλον της κινέζικης πολιτικής περνάει από τις ασφάλειες, από τις ασφαλίσεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είπατε ότι τα άρθρα 37, 38 και 39 του κανονισμού 1305 είναι ενδιαφέροντα γιατί προτείνουν να βοηθήσουν τις ασφαλίσεις αλλά να βοηθήσουν και τα βιβλία κεφάλαια. Οπότε δεν θα περάσουμε αποκλειστικά στις ασφαλίσεις ως τρόπο διαχείρισης του κινδύνου, όπως ε, υπενηχθήκατε με τις ερωτήσεις. Η έννοια των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο που στηρίζεται στην ε, αλληλεγγύη μεταξύ των γεωργών. Και εκεί θα πρέπει να αναζητήσουμε τις λύσεις για το μέλλον. Δεν θα βρούμε εκείνη λύση ε, για τα απορροκυπευτικά ή το γαλακτοκομικό τομέα ή την ίδια λύση για το βορρά και το νότο. Είναι τόσο διαφορετικές οι καταστάσεις και τόσο πολλές ιδιαιτερότητες που δεν μπορούμε να έχουμε ένα γενικό σύστημα που θα ισχύει για όλους. Τώρα, αν θα περάσουμε από τις άμεσες ενισχύσεις σε ένα σύστημα ασφαλιών που θα οδηγεί στον πλουτισμό των ασφαλιστικών εταιριών, όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι οι άμεσες ενισχύσεις θα οδηγήσουν σε διέξοδο. Πολλοί είναι υπέρ των άμεσων ενισχύσεων, αλλά άλλοι ε, είναι κατά. Είναι αφιλεγόμενες οι άμεσες ενισχύσεις. Και το θέμα δεν είναι ότι σχετίζονται με τους παράγοντες της παραγωγής, το, την αξία της γης και ούτω καθεξής. Αλλά όπως είπε και ο Λιθουανός Ευρωβουλευτής, η αξία των άμεσων ενισχύσεων περνά και στη διανομή. Και όσο περισσότερες ενισχύσεις δίνονται στη γεωργία, τόσο πιο εύκολο είναι στα μεγάλα σούπερ μάρκετ να απομυζήσουν τους γεωργούς. Οπότε οι άμεσες ενισχύσεις δεν επιλύουν το θέμα του βιοπορισμού των μικρών καλλιεργητών, των μικρών γεωργών. Εκτός και αν γίνει μια διαφοροποίηση των άμεσων ενισχύσεων για τους ε, γεωργούς μικρής ε, κλίμακος. Στη Ρουμανία έχουμε πολλούς μικρούς καλλιεργητές που δεν ε, υπησέρχονται στο περίπλοκο σύστημα των αμοιβαίων κεφαλαίων και ούτω καθεξής. Ούτε και τις άμεσες ενισχύσεις που είναι και αυτές σε ένα περίπλοκο σύστημα. Ίσως για τους μικρούς καλλιεργητές Θέλουμε ένα πιο απλό και άμεσο σύστημα. Για τη μεγάλη όμως πλειοψηφία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι σύγχρονες και στραμμένες προς το μέλλον, θα πρέπει να βρούμε κάποια συστήματα για το μέλλον. Δεν είναι ότι θα πρέπει να ε, μοιραστούν όλοι ένα περιορισμέ, μια περιορισμένη πίτα άμεσων ενισχύσεων είτε ανάντι είτε κατάντι. Θα πρέπει με το διαθέσιμα κονδύλια να αναπτύξουμε σταδιακά ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνων, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες επενδύσεις και για τις μεγάλες καλλιέργειες, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μερικοί μεγάλοι καλλιεργητές ε, έχουν και μαζικές παραγωγές. Στη Ρουμανία γνωρίζω ένα συνεταιρισμό που έχει 20.000 εκτάρια. Ε, έναν μάλλον ε, μεγαλοκαλλιεργητή που δεν ανήκει σε συνεταιρισμό. Επίσης έχουμε δίπλα αυτές τις τεράστιες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μικρές εκμεταλλεύσεις ενός εκταρίου. Δεν μπορεί να ισχύει το ίδιο σύστημα για τις διαφορετικές καταστάσεις. Μερικές εκμεταλλεύσεις και μερικοί γεωργοί θα επενδύσουν για να έχουν μαζική παραγωγή με χαμηλό κόστος. Άλλοι θα κάνουν πιο πρωτότυπες επενδύσεις, ώστε να κάνουν άμεσα τις παραδόσεις τους στους καταναλωτές με άμεσες πωλήσει. Και γι' αυτό για το μέλλον είναι ενδιαφέροντα και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων γιατί ε, διανοίγονται ευκαιρίες για όλους και δεν μοιραζόμαστε ένα περιορισμένο, ε, μια περιορισμένη πίτα αλλά την διευρύνουμε. Επίσης υπάρχουν μεγάλες τεχνικές διαφορές μεταξύ των ασφαλιστικών συστημάτων στην Αμερική και εδώ. Οι κλασικές ε, ασφαλιστικές επιχειρήσεις εγγυώνται τις, τις απώλειες σε ένα εγγυημένο κεφάλαιο. Οπότε, αν έχουμε διαδοχικές καταστροφές, οι ασφάλειες πληρώνουν σε συνεχόμενα έτη. δεν ισχύει το ίδιο για τα αμοιβαία κεφάλαια. Τα αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να πληρώσουν μόνο εφόσον έχουν κεφάλαιο. Οπότε, αν έχουν ένα ανεπιθύμητο συμβάν, μια θεμενία, θα πρέπει να το σκεφτούν και οι μέτοχοι, οι γεωργοί θα πούνε να κρατήσουμε και ένα απόθεμα, ένα αποθεματικό. Γιατί αν του χρόνου έχουμε νέα θεομηνία ή άλλη καταστροφή ή κάπου αλλού που καλύπτεται από το αμοιβαίο κεφάλαιο, θα χρειαστούμε και του χρόνου κεφάλαια. Και αυτή η σκέψη και η, η φρόνιμη διαχείριση του κινδύνου μας επιτρέπει να βάλουμε τις βάσεις για να δούμε το ύψος της αποζημίωσης. Οπότε ισχύει εδώ η τοπική αλληλεγγύη με ελάχιστη βοήθεια από τις δημόσιες αρχές. Για τις ε, καταστροφές έχουμε 30% μόνο του, της απώλειας παραγωγής που κινητοποιεί τα κρατικά κονδύλια. Για τις μικρές απώλειες δεν έχουμε βοήθεια. Ενώ οι άμεσες ενισχύσεις δεν λαμβάνουν κάτι τέτοιο υπόψη. Δίνουν ε, χρήματα ψηλώ ανάλογα με ιστορικά κριτήρια αναφοράς. Είτε με βάση την καλλιέργεια είτε με βάση τη χώρα. Ενώ έχουμε συστήματα εμεί που θα πρέπει να συνδυάσουν τα μηδέα κεφάλαια και την αλληλεγγύη με ένα σύστημα διαχείριση κινδύνων. Και αυτό επιζητούν και οι γεωργοί. Επίσης, Τα 10% από τις άμεσες ενισχύσεις δεν θα τροφοδοτήσουν τις ασφαλίσεις. Καθόλου. Δεν πρότεινα κάτι τέτοιο. Και το γεγονός ότι οι πανεπιστημιακοί κάνουν κάποιους υπολογισμούς ε, αναλογιστικούς ή όπως είπα και για τη Ρουμανία κάνουν δειγματοληψίες αντιπροσωπευτικές ε, για να απολογιστούν οι κίνδυνοι, θα πρέπει κάπως να προσδιορίσουμε τις τοπικές απώλειες μετά από μια θεομηνία, από μια καταστροφή. Χρειάζονται γι' αυτό στατιστικολόγοι. Δεν θέλω ε, έτσι να τροφοδοτήσουμε τα, τα πανεπιστήμια, αλλά θα πρέπει να γίνει με σωστή ανάλυση των ε, δεδομένων. Το είπε και ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στι ΗΠΑ υπάρχουν στοιχεία για τι ιστορικέ αποδόσει τη κάθε εκμετάλλευση. Ε, οπότε έτσι με τις βάσεις δεδομένων περιορίζονται οι απάτε. Εμείς τι κάνουμε για να προχωρήσουμε. Εμείς απλώ μετράμε τα στρέμματα και ε, μοιράζουμε χρήματα με βάση τεχνικά στοιχεία. Θα πρέπει με τη γνώση να προχωρήσουμε. Επαναλαμβάνω, δεν είπα να πάρουμε τα χρήματα από τις άμεσες ενισχύσεις και να τα δώσουμε στις ασφαλιστικές ή στα πανεπιστήμια. Επουδενή. Επίσης, τέθηκε μια ερώτηση για τη διαφοροποίηση μεταξύ των μικρών καλλιεργητών που ίσως χρειαστούν μια παρακολούθηση για τις άμεσες ενισχύσεις σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες που έχουν ε, ένα τέτοιο σύστημα ανεπτυγμένο και είναι έτοιμες ήδη να λειτουργήσουν. Επίσης μιλήσαμε για, το, για την ισχύ της αγοράς και τα χρήματα που καρπώνονται οι μεσάζοντες και τα σούπερ μάρκετ. Οπότε φεύγουν τα χρήματα από τον παραγωγό. Δεν είναι αποτελεσματικές εδώ οι άμεσες ενισχύσεις. Τώρα, για τα κρατικά κονδύλια που πηγαίνουν προς τον Γεωργό για ένα δολάριο που επενδύει ο Γεωργός στις Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνει δύο. Οπότε οι αμερικανικές ασφαλίσεις μεταφέρουν τα κονδύλια και τον υπολογισμό προς τους γεωργούς. Πολύ σημαντική βοήθεια λοιπόν για τους γεωργούς. Οι υπολογισμοί βέβαια είναι ιδιαίτερα περίπλοκοι το ευρωπαϊκό σύστημα όπως προβλέπεται στα κείμενα μια επιδότηση του ύψους του 65% των αμοιβαίων κεφαλαίων δηλαδή αν Γεωργιός ε, ε, επενδύσει 3, 3,5 ή 35 ευρώ στα 100 και υπάρξει μετά μια απώλεια θα πάρει 100 γιατί 65 θα είναι η δημόσια ενίσχυση και ο Γιώργος ε, μπορεί να πει ότι βάζω ένα, παίρνω το διπλό. Τι συμπέρασμα προκύπτει από αυτό. Ποιος ε, χρηματο, χρηματοδοτεί αυτό το σύστημα. Ποιος προσθέτει, ποιος συμπληρώνει ώστε ο Γιώργος να πάρει το διπλάσιο από αυτό που επενδύει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. επαναλαμβάνω. Αυτή την ε, συνοπτική μου επιχειρηματολογία που είναι και κάπως δημοσιογραφική. Μπορεί να αναφερθεί έτσι. Στο ευρωπαϊκό κείμενο. Αν χάσει κανείς πάνω από το 30% της οδιάς του, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο άρθρου 38 θα του δώσει ας πούμε 100 ευρώ και από αυτά τα 100 ευρώ ο Γιωργός θα έχει πληρώσει ασφάλιστρα 35%, 35 ε, ευρώ και τα 65 ευρώ θα είναι δημόσια ενίσχυση. 75% η ένωση του ποσού αυτού και 25% τα κράτη-μέλη. 35 δίνει ο παραγωγός, παίρνει 100 αποζημίωση. Απλός υπολογισμό. Βάζω 3, παίρνω 6. Άρα παίρνω το διπλάσιο. Βέβαια είναι απλουστευμένοι, υπεραπλουστευμένοι αυτοί οι υπολογισμοί. Δεν αντανακλούν πώ ακριβώ λειτουργεί το σύστημα. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε πώ χρησιμοποιούμε του αριθμού. Γιατί κατόπιν ε, το παίρνει μία πηγή από την άλλη και δεν είναι και πολύ ακριβής. Άλλο πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση για το βραχή και το μακροπρόθεσμο. Τι να κάνουμε. Με βάση την υπάρχουσα κατάσταση. Κοιτάξτε, το πρόβλημα με τη διαχείριση κινδύνων είναι ότι χρειάζεται πλούσια πείρα. Αυτά τα συστήματα δεν μπορούμε να τα επινοήσουμε από τη μια μέρα στην άλλη και να πούμε, ε, ας κάνουμε αυτό και μια χαρά θα τα πάει. Όχι, πρέπει να υπάρξει μια περίοδος μαθητείας, μαθαίνει κανείς από τα λάθη του, προχωρεί, δημιουργεί βάση δεδομένων, ελέγχει τα στοιχεία του. Αν κάνουμε, θέλουμε να βασιστούμε στο παρελθόν της παραγωγής, πρέπει να έχουμε στοιχεία για το παρελθόν της παραγωγής. Και μετά πρέπει να υπάρξουν και μεταβατικά συστήματα. Άρα, από τη μια μέρα στην άλλη, δεν θα περάσουμε από ένα σύστημα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πρέπει να σκεφτούμε και τις μεταβατικές φάσεις. Αλλά και το στόχο μας. Για να προχωρήσουμε λοιπόν να βοηθήσουμε αυτούς που είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν, που θα λάβουν υπόψη τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά και που θα ζητήσουν να δημιουργηθούν αμοιβαία κεφάλαια με ειδικού όρους, για παράδειγμα για τα απορκυπευτικά, να αφήσουμε από κάτω προς τα πάνω να υπάρξουν οι εξελίξεις, να τους στηρίξουμε, να υπάρξει ανταλλαγή πείρας από τη μια χώρα στην άλλη, ούτως ώστε όποιες ιδέες προκύψουν να συζητηθούν μεταξύ όλων και να ε, βελτιωθούν. Όχι λοιπόν επανάσταση, εξέλιξη. Δεν θα πάμε το 1,3% στο 10% έτσι με τη μία. Θα έχετε χρόνο να εξηγήσετε στους Γεωργούς τι γίνεται και γιατί και γιατί είναι προς το συμφέρον τους. Δεν χρειάζεται να πούμε θα σας πάρουμε τα λεφτά. Όχι, αύριο. Όχι, όλα αυτά θα γίνουν σταδιακά. Τέλος. Αν και νομίζω ότι απάντησα σε όλα. Πολύ με ενδιαφέραν και πολύ ενδιαφέροντα βρήκα και αυτά που λέει η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για τα δεδομένα. Ναι, βεβαίως, πρέπει να επενδύσουμε στα στοιχεία, στη γνώση. Όχι, να μην μοιράσουμε την πίτα. Θέλω μια μεγάλο κομμάτι εγώ, άρα θα πας λιγότερο εσύ. Όχι, να φτιάξουμε μια μεγαλύτερη. Να ε, ε, αναπτύξουμε την ικανότητα των γεωργών να κάνουν τις σωστές επενδύσεις. Και ο γεωργός τελικά θα ωφεληθεί. Ελπίζω να απάντησα σε όλα. Γενικά. Και ελπίζω να ε, έδωσα απαντήσεις σε αυτούς που έθεσαν τα ερωτήματα. Σίγουρα, αν είχαμε περισσότερο χρόνο, θα υπέβαλαν και άλλες ερωτήσεις, συνάδελφοι, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας είναι μετρημένος. Και η κοινή γεωρική πολιτική σίγουρα βρίσκεται σε εξελικτική πορεία. Και όλο και περισσότερο μιλούμε για την εφαρμογή και κάποιων χρηματοοικονομικών μέσων. Σίγουρα λοιπόν θα πρέπει να εξετάσουμε αν αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα θα είναι δημόσια, κοινοτικά, γιατί χρειάζονται και τέτοιου είδου μέτρα μέσα θα πρέπει να είναι ελαστικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε προγραμματισμό, γιατί η κατάσταση μεταβάλλεται. Μερικές φορές χρειάζονται περισσότερα, τέτοια μέσα άλλες φορές λιγότερα, ανάλογα με τις συνθήκες. Οπότε θα πρέπει να γίνει μια εξατομίκευση των ενισχύσεων και της ασφάλισης των ε, γεωργών. Δεν υπάρχει, είπατε δεν είναι νέο σύστημα. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικές ενισχύσεις, αλλά ταυτόχρονα να αποφύγουμε και τις απάτες. Και το σύστημα αυτό χρειάζεται χρόνια για να αναπτυχθεί. Αλλά νομίζω ότι προς αυτή την πορεία θα κινηθεί η εξέλιξη στην κοινή γεωργική μας πολιτική. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Νομίζω ότι οι προτάσεις σας θα τροφοδοτήσουν και τις συζητήσεις και θα μας εμπνεύσουν και χαράζουν και μία πορεία για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Δυστυχώς το πρόγραμμα μας είναι πολύ γεμάτο και πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Λυπούμε που δεν είχαμε περισσότερο χρόνο για να αφιερώσουμε στις ερωτήσεις και στη συζήτηση, γιατί πραγματικά η παρουσίαση της μελέτης σας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστούμε λοιπόν τον καθηγητή και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι βουλευτές της Επιτροπής μας ε, επαρελειμμένως επέκριναν το νέο σύστημα των άμεσων ενισχύσεων εξαιτίας της περιπλοκότητάς του. Και ο προηγούμενος καλεσμένος μας εν μέρη έθιξε το θέμα αυτό. Είπε για παράδειγμα ότι οι άμεσες ενισχύσεις βρίσκονται σε ένα διέξοδο. Ότι το σύστημα αυτό έχει προσκρούσει σε διέξοδο θα πρέπει να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για την εφαρμογή του συστήματος και γι' αυτό ε, συζητήσαμε και το θέμα με τον Επίτροπο Χόγκαν και σήμερα έχουμε τον Διευθυντή της ε, Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη, τον κύριο Πιέρ Μπασκού, που θα μας κάνει μια ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του συστήματος άμεσων ενισχύσεων σε όλα τα κράτη-μέλη. Δίνω το λόγο λοιπόν στον κύριο Μπασκού. Σας ακούμε κύριε Μπασκού. Thank you very much, I would like to do in this presentation for around, I think, 15 minutes. Γύρω στο 1 τέταρτο θα διαρκέσει η παρουσίασή μου. Αυτό μου είπε ο πρόεδρος ότι δικαιούμαι. Και θα ήθελα να σας κάνω μια γενική επισκόπηση του νέου συστήματος άμεσων ενισχύσεων και το πώς θα εφαρμοστεί αυτό επί τη βάση της, των κοινοποιήσεων που στέλνουν τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μάλιστα ε, είναι πολύ επίκαιρη αυτή η συζήτηση γιατί λίγη προθεσμία της κοινοποίηση. Ε, αναμένονται κάποιες ε, μικρές αλλαγές, αλλά νομίζω ότι η επισκόπηση που θα σας κάνω είναι σχετικά πλήρης για το μέλλον των άμεσων ενισχύσεων και το νέο κανονιστικό πλαίσιο που ξεκινά να εφαρμόζεται από το ξεκίνημα του έτους. Οπότε οι άμεσες πληρωμές έχουν σημαντικό ρόλο και πρέπει να έχουμε μια συνθετική εικόνα για το πώς εφαρμόζονται οι απευθείας ενισχύσεις και πώς θα κερδίσει ο Γεωργός στο μέλλον. Θα ξεκινήσω την παρουσίαση αυτή με υπενθυμίζοντας τις βάσεις ε, της διαδικασίας και μετά θα σταθώ στα βασικά στοιχεία των αλογών τονίζοντας θέματα που αφορούν το greening και άλλα κομμάτια των απευθείας ενισχύσεων. Πρώτον, να Μία ενημέρωση για τις ε, πολιτικές ε, των κρατών μελών που υιοθετήθηκαν στις 23 Ιανουαρίου, πριν από λίγες εβδομάδες δηλαδή. Ε, η έκθεση, της, η αναφορά μάλλον της κοινοποίησης προς τα κάτι μέλη δεν συνιστά έγκριση από την Επιτροπή αυτών των κοινοποιήσεων. Δύο λόγια τώρα για τη διαδικασία προς υπονθύμηση. Σας θυμίζω, αλλά το ξέρει το ξέρετε, η Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει τις κοινοποιήσεις των κατων μελών. Παραμένουν οι μόνοι υπεύθυνοι δι' αποφάσεων πολιτικών που λαμβάνονται και απλά κοινοποιούν τις αποφάσεις του στην Επιτροπή. Δύο εξαιρεσει υπάρχουν στο Γενικό Κανόνα. Πρώτον, εθελοντική υποστήριξη όταν τα κράτη-μέλη δώσουν πάνω από 13-15% στο voluntary capping support συνδεδεμένη υποστήριξη και σε περιπτώσεις ισοδύναμο ε, greening, μια διαδικασία αξιολόγησης όπου η Επιτροπή πρέπει με την απόφαση να ενημερώνει τα κράτη-μέλη που έδωσε την κοινοποίηση για το μηχανισμό ε, χρησιμοποίησης της ε, διαδικασίας greening ή την απόρριψη. Άρα η Επιτροπή δεν χρειάζεται να εγκρίνει να απορρίψει την κοινοποίηση. Γι' αυτό οι περισσότερες ανταλλαγές απόψεων που, έχουν, ε, που τα κράτη-μέλη τους τελευταίους 7-8 μήνες ε, ασχολήθηκαν με την αξιολόγηση της ε, πληρότητας και της συνέπειας της κοινοποίησης. Ενώ ταυτόχρονα συζητήσαμε με τα κράτη-μέλη το πώ θα εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση της κοινοποίηση από πλευρά και των μελών με το νέο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις απευθεία ενισχύσει. Είχαμε πολλές διμερείς ε, επαφές, πάνω από 100 συναντήσεις με εκπροσώπου της διοίκηση, Υπουργεία, ε, οργανισμούς πληρωμών, με εμπλεκόμενου φορεί. Είχαμε μια εντατική ανταλλαγή απόψεων με τα κράτη-μέλη, τους τελευταίους οκτώ μήνες σε σχέση με τις ε, κοινοποιήσεις αυτές. Προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε μία σύνοψη των βασικών αποφάσεων πολιτικής. Θα σταθώ ωστόσο για την υπόλοιπη παρουσίασή μου σε αυτά παρουσιάζοντας τις αποφάσεις των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την ευελιξία μεταξύ πυλώνων, την ε, μείωση των πληρωμών, τις επιλογές που αφορούν στα βασικά προγράμματα πληρωμής, το εφελούσιο συνδεδεμένη, την εθελούσια συνδεδεμένη υποστήριξη και του τομεί που, που καλύπτονται. Τώρα, η ευελιξία μεταξύ πυλώνων. Τα κράτη-μέλη έχουν να μεταφέρουν ποσά από μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα ή δεύτερου και πρώτου πυλώνα. Όπως βλέπετε από τον πίνακα εδώ, μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα, τα 11 κράτη-μέλη αποφάσισαν να γίνει μεταβίβαση χρηματοοικονομικών ποσών στο δεύτερο πυλώνα, συνολικά 6,4 δις ευρώ. Ταυτόχρονα 5 κράτη αποφάσισαν να περάσουν πόρους από τον δεύτερο στον πρώτο πυλώνα, συνολικού ποσού 3,4 δις ευρώ. Αυτές είναι οι χώρες που βλέπετε στο κάτω μέρος του πίνακα. Οι μεταφορές, το καθαρό ποσό μεταφοράς μεταξύ πρώτης, δεύτερης και δεύτερης πρώτης είναι από τον πρώτο προς το δεύτερο καθαρό ποσό 3 δις τα επόμενα 6 χρόνια. Μισό δις κάθε χρόνο δηλαδή. Στον πίνακα αυτό προσπαθούμε να συνοψίσουμε τις βασικές αποφάσεις πολιτικής των κρατών μερών στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου συστήματος άμεσων ενισχύσεων. Αν δείτε τον πίνακα, θα διαβάσετε τον πίνακα, θα δείτε ότι τα 10 κρατημέλη που εφαρμόζαν το σύστημα μέχρι το 2014, συνεχίσουν να το κάνουν αυτό, το SAPS δηλαδή, μέχρι το 2020. Έξι χώρες έχουν αποφασίσει να, περιο... να περιφερειοποιήσουν το βασικό σύστημα πληρωμών τους ε, χρησιμοποιώντας το άρθρο 23 Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Φιλανδία και Βρετανία. Οκτώ χώρες ανακοίνωσαν στην Επιτροπή ότι εισήγαγαν ένα σύστημα αναδιανομητικών πληρωμών χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα παροχής επιπλέον ε, απευθείας ενισχύσεων στις μικρές και μεσαίες ε, εκμεταλλεύσεις και από τα 8, από τα 8 κράτη 6 χρησιμοποίησαν τη δυνατότητα των πληρωμών αυτών και την μη υποχρεωτική μείωση των μηχανισμών πληρωμής, τη δυνατότητα δηλαδή που της παρέχεται αυτή. Μία μόνο χώρα χρησιμοποίησε την δυνατότητα να δώσει από δεσμευμένες ε, πληρωμές ε, η Δανία ενώ 27 από τις 28 χώρες, με την εξαίρεση της Γερμανίας, 27 ανακοίνωσαν ότι θα έχουν την εθελούσια συνδεδεμένη υποστήριξη. Θα επανέλθω σε αυτό. 15 χώρες τώρα αποφάσισαν να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα μικρών, μικρής γεωργίας, 15 από τις 28 και από τις 15 αυτές δύο αποφάσισαν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα αυτό με εφάπαξ ποσό. Όλες οι άλλες χώρες έδωσαν στους μικρούς γεωργούς συγκεκριμένο ποσό που, βάση, που οφείλεται βάσει του συστήματος είτε για το 2015 είτε το μερίδιο μέχρι το 2020. Αυτή είναι η γενική εικόνα των αποφάσεων πολιτικής. Αν δείτε το πώς οι αποφάσεις αυτές μεταφέρονται σε δημοσιονομικό κόστος για κάθε επίπεδο απευθείας ενίσχυσης ανά κράτος μέλος, Βλέπετε στον πίνακα εδώ ότι 30% του εθνικού, του εθνικού χαρτοφυλακίου πηγαίνει για τις πράσινες εθελούσιες πληρωμές. Η εθελούσια συνδεδεμένη υποστήριξη ποικίλει από χώρα σε χώρα, αλλά κατά μέσο όρο είναι γύρω στο 10% του συνολικού ποσού των απευθείας ενισχύσεων που παρέχονται στους γεωργούς. Βλέποντας τώρα τι έχει μείνει στην ουσία, βασικό πρόγραμμα πληρωμών και SAPS, που είναι τα, οι παλιέ αποσυνδεδεμένε πληρωμέ. βλέπουμε ότι σε μέσο όρο στην Ένωση αντιπροσωπεύουν το 55% του συνολικού εθνικού ε, χαρτοφυλακίου. Οι αποσυνδεδεμένες αυτές πληρωμές ε, κατά μέσο όρο είναι 55 όπως σας είπα, 20% Μάλτα, 38% στη Λιθουανία, ενώ η Ιρλανδία, η, Ολλανδία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία έχουν γύρω στο 68%. Υπάρχει δηλαδή μια αναδιανομή των συνολικών κονδυλίων μεταξύ διαφόρων επιπέδων και βλέπουμε ότι τα κράτη που επέλεξαν την εφαρμογή αναδιανομητικών πληρωμών το ποσοστό που έδωσαν για αυτές τις πληρωμές ανέχεται από 5 έως 15%. Αν δείτε τώρα την μείωση των μηχανισμών, τον μηχανισμό μείωση των πληρωμών, βλέπετε ότι 9 κράτη-μέλη αποφάσισαν να θέσουν ανώτατο όριο στη μείωση του BPS, ανώτατο όριο 150, μεταξύ 150 και 600.000 ευρώ, Βλέπετε τα διάφορα επίπεδα ανά κράτος μέλος. 15 κράτη-μέλη θα εφαρμόσουν μόλις την υποχρεωτική ελάχιστη πληρωμή, μείωση πληρωμής 5% για τα ποσά άνω των 150.000 ευρώ, ενώ ο μηχανισμός αυτός μείωσης των πληρωμών συνολικά καλύπτει 558 εκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 5 για τα επόμενα 5 χρόνια. Λίγο πάνω από 100 εκατομμύρια το χρόνο. Πολύ χαμηλό ποσό αν το συγκρίνουμε με τον, επίσημο, με τον ετήσιο χρήμα προϋπολογισμό ε, που σε ετήσια βάση είναι γύρω στα 48 δισεκατομμύρια. Τώρα, το BPS, το βασικό, το, βασικό πρόγραμμα πληρωμών, αν δείτε πώς εφαρμόζεται η εσωτερική σύγκληση μεταξύ των οκτώ κρατών μελών που εφαρμόζουν το BPS, 7 έχουν πετύχει μια μορφή εθνικού ή ε, περιφερειακού καταποκοπή ποσού, η Γερμανία, η Κορσική στη Γαλλία, η Κωσική στη γαλλια η μαλτα και η Αγγλία μόνο στη Βρετανία το 2015, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φιλανδία, η Σκοτία και η Ουαλία το 2019 και η Σουηδία θα φτάσει το καταποκοπή ποσό το 2020. Όλα τα άλλα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν το BPS επέλεξαν μια μερική σύγκληση. Οι περισσότερες δε χώρες 11 συγκεκριμένα επέλεξαν τη δυνατότητα περιορισμού της μείωσης της αξίας του βασικού συστήματος πληρωμής παν, 30% πάνω από το μέσο όρο. Τώρα, το VPS, το Voluntary Coupled Support, όπως σας είπα, κατά μέσο όρο στην Ένωση, το 10% του συνολικού εθνικού πακέτου πηγαίνει στην εθελούσια ε, συνδεδεμένη υποστήριξη. Όπως βλέπετε, από αυτό τον πίνακα εννέα χώρες αφιερώνουν ε, λιγότερο από 8% στο VCS και 11 κράτη-μέλη έχουν ε, ανέβει στο μέγιστο επιτρεπόμενο 13% ή και 15% αν πρόκειται για σοδιές πρωτεϊνούχες. Τρία κράτη-μέλη θα χρειαστεί να λάβουν ε, έγκριση από την Κομισιόν γιατί υπερέβησαν το 15% Βέλγιο, Φιλανδία, Πορτογαλία. Και η Μάλτα δεν αναφέρεται, είναι ειδική περίπτωση, πάει το 57% στο VCS και η Γερμανία που είναι 0%. Να δούμε τώρα τους διάφορους τομείς που αφορώνται από το VCS. Συνολικά σε ενωσιακό επίπεδο είναι 259 τέτοια μέτρα, μεγάλος αριθμός, είναι νομίζω και όμως ε, ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ ε, κλάδων και χωρών. Να δούμε τώρα την ε, απόλυτη αξία. Πρώτα απ' όλα, κύριος χρήστης είναι ο τομέας ε, των ε, ζώων. Αυτοί και τα επόμενα χρόνια θα λάβουν τη μερίδα του λέοντος γιατί 42% πάει στο βόλιο, 20% στον γαλακτοκομικό τομέα, 12% στα εγω... προ... πρόβατα. Μεγάλο ποσοστό λοιπόν είναι όπως βλέπουμε εδώ το 2015 στον ε, τομέα των ζώων. Θα υπάρξει μια ποικιλία μέχρι το 2020, αλλά συνολικά για τα επόμενα 5-6 χρόνια θα είναι σχετικά σταθερό το ποσοστό. Τώρα για να δούμε τώρα τη ρήτρα για τον ενεργό γεωργό. Δεν μπορεί κανείς να ζητήσει να ε, αμυφθεί αν εργάζεται κυρίως σε ορισμένους τομείς που αναφέρονται σε ένα αρνητικό κατάλογο Βλέπουμε ότι 8 κράτη-μέλη προσέθεσαν και κάποιες δραστηριότητες σε αυτόν τον ε, αρνητικό κατάλογο. Βλέπετε τις χώρες εδώ. Έχουν προσθέσει διάφορες αρνητικές δραστηριότητες, για παράδειγμα διαχείριση ε, των δασών, ορυχεία και τράπεζες, έξι κράτη-μέλη αποφάσισαν να δώσουν αυτές χρηματοδοτήσεις σε όλους εφόσον έχουν σημαντικό τμήμα της δραστηριότητάς τους να συνδέεται στην, ε, που να είναι γεωργική ή αν η δραστηριότητά τους συνδέεται με τη γεωργία. Και υπάρχουν και διάφορα κατόφλια εξαιρέσεων. Να δούμε τώρα το πρασίνισμα που έχει συζητηθεί τόσο πολύ την τελευταία τετραετία εδώ συνοψίζουμε μερικές βασικές αποφάσεις που σχετίζονται με το πρασίνισμα. Αριστερά βλέπετε πέντε κράτη-μέλη μας έχουν ενημερώσει για τους ισοδύναμους μηχανισμούς πρασινίσματος. Τέσσερα κράτη-μέλη αποφάσισαν να εφαρμόσουν σε περιφερειακό επίπεδο τις μόνιμες αναλογίες Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο και Ηνωμένο Βασίλειο. Δύο κράτη-μέλη αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν τους ε, τομείς ε, οικολογικής εστίασης και δεξιά τη βλέπετε τέσσερις από τις πέντε χώρες που μπορούσαν να ωφεληθούν από την ε, εξαίρεση για τα δάση Τέσσερι αποφάσισαν να τι εφαρμόσουν αυτέ τι εξαιρέσει. Εστονία, Φιλανδία, Λετωνία και Σουηδία. Μόνο η Σλοβενία αποφάσισε να μην εφαρμόσει αυτή την εξαίρεση για τα δάση. Ποιε είναι οι τρει υποχρεώσει πρασινίσματο. Είδαμε ποιε χώρε μέλη μα ενημέρωσαν μέσω συστημάτων πιστοποίηση ενώ τρία κράτη-μέλη αξιοποίησαν το δεύτερο πυλώνα και η κύρια πρακτική για το πρασίνισμα είναι η υποχρέωση πιστοποίησης. -μέλη, μόνο δύο κράτη-μέλη ε, αξιοποίησαν άλλες δυνατότητες. Αν δούμε τώρα τις υποχρεώσεις των οικολογικών περιφερειών ε, εστίασης. Διαπιστώνουμε εννιά διαφορετικά είδη τοποθεσιών. Οπότε τα κράτη-μέλη αποδεικνύεται ότι διαφορετικά έχουν αντιμετωπίσει την κατάσταση. Έξι κράτη-μέλη αποφάσισαν να περιορίσουν τους τομείς αυτούς. Βλέπετε ποιες χώρες είναι σε αυτή τη διαφάνεια και 13 κράτη-μέλη αποφάσισαν να προσφέρουν πολλές δυνατότητες αυτού του EFA στους γεωργούς. Αν δείτε τι κατηγορίες EFA επελέγησαν, βλέπετε εδώ στο κάτω μέρος, ποια κράτη-μέλη που μας ενημέρωσαν γιατί είδος EFA διάλεξαν. Για παράδειγμα, οι δύο τύποι που αξιοποιούνται περισσότερο είναι οι σοδιές που δεσμεύουν το άζωτο και οι ε, σύντομες εναλλαγές καλλιεργιών. Τώρα δούμε τα χαρακτηριστικά των τοποθεσιών. Έχουμε 9 διαφορετικές ε, δυνατότητες επιλογής χαρακτηριστικών τοποθεσιών και βλέπουμε τι επιλογές έχουν γίνει στα διάφορα κράτη-μέλη. Ορισμένοι βάζουν ομάδες ε, δέντρων, άλλοι προτιμούν ε, διαδρόμους μεταξύ των χωραφιών, άλλοι σειρά δέντρων. Ο καθένας επιλέγει αυτό που είναι πιο κατάλληλο. Βλέπουμε λοιπόν τι διαφορετικές επιλογές έχουν γίνει για αυτό το είδος ε, EFA, περιοχών οικολογικής εστίασης δηλαδή. Τα κράτη-μέλη έχουν δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν μόνο τους κανόνες στο άρθρο 45 ή, τις, ε, ή τους κανόνες της κατεξοδότηση πράξης ή να αξιοποιήσουν τους κανόνες που αφορούν την πολλαπλή συμμόρφωση Βλέπουμε ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη επέλεξαν να επιτρέψουν και τους δύο ορισμούς που υπάρχουν και με βάση το άρθρο δηλαδή 45 και με βάση την πολλαπλή συμμόρφωση. Και η τελευταία διαφάνεια αφορά τις υποχρεώσεις για μόνιμους χορτοτόπους την υποχρέωση που έχουν δηλαδή τα κράτη-μέλη να ενημερώσουν για ποιες τέτοιες ε, περιοχές λιμονών έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν. Οκτώ κράτη-μέλη αποφάσισαν όλοι οι λιμόνες τους να μπουν στο Natura 2000 και να θεωρούνται λοιπόν οικολογικά ευαίσθητοι μόνιμοι λιμόνες. Πέντε κράτη-μέλη επέλεξαν να συμπεριλάβουν μεταξύ 50 και 100 και για τα υπόλοιπα θα πρέπει να δούμε. Τελευταίο που θέλω να αναφέρω για αυτή την υποχρέωση για τους μόνιμους λιμόνες, τέσσερα κράτη-μέλη αποφάσισαν να καθορίσουν τέτοιες περιοχές πολύ ε, με πολύ πιο αυστηρές προδιαγραφές. Εκτός των περιοχών του Natura 2000, η Τσεχική Δημοκρατία, το Λουξεμβούργο, η Λετωνία και η Ουαλία. Αυτά θέλησα να κάνω μια αναλυτική επισκόπηση. Φυσικά, αν θέλετε, μπορούμε να πάμε και σε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες και ελπίζω αυτή η παρουσίαση να σας έχει επιτρέψει να καταλάβετε πώς θα εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες ε, στα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Σίγουρα μας ενδιαφέρουν και οι λεπτομέρειες, γι' αυτό και θα θέσουμε σχετικές ερωτήσεις. Κύριε Ντες, είχα στοιχηματίσει ότι εσείς πρώτος θα ζητήσετε το λόγο. Τον έχετε λοιπόν. Ευχαριστώ Πρόεδρο. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Συνέβη αυτό ακριβώς που φοβόμασταν. Όλο και λιγότερο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε μια κοινή γεωρική πολιτική. Μετά τη μεταρρύθμιση οι διαφορές στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες έχουν ε, μεγαλώσει πάρα πολύ. Πολύ περισσότερο από ό,τι ήσαν πριν από 20 χρόνια. Αυτό θα μας οδηγήσει σε μεγάλες τρευλώσεις του ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Αυτό που κυρίως με λυπεί είναι ότι αυτές οι διαφορές μέχρι το 2019-2020 θα διατηρηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ποια είναι η κατάσταση στη Γερμανία. Στη Γερμανία η περιοχή μου είναι σε μειονεκτική θέση. Σε όλες τις περιοχές της Γερμανίας το 19 ανά θα πρέπει να πληρώνουμε το ίδιο ποσό. Δηλαδή η Ρινανία, ε, Βεσφαλία, όπου ε, έλαβαν ε, λιγότερες πληρωμές λόγω καλύτερης οδιάς, θα πρέπει να λαμβάνουν τις ίδιες πληρωμές. Αυτό νομίζω ότι είναι δίκαιο διότι βεβαίως στις πιο μειονεκτικές περιοχές είναι πολύ δύσκολες ε, οι συνθήκες. Αυτό που επιτύχαμε είναι στη Γερμανία περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ πέρασε από την ε, καλλιέργεια εδαφών στην ε, χρηματοδότηση των χορτοτόπων, των λιμονών. Αυτό νομίζω είναι πολύ καλό. Στη Γερμανία μπορούμε να επιδοτήσουμε μέχρι και 46 εκτάρια. Και πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διαφορές μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων και αν υπάρχουν να είναι προς όφελος των μικροτέρων εκμεταλλεύσεων. Πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουμε το θέμα αυτό και στα πλαίσια περαιτέρω μεταρρυθμίσεων. Γιατί δεν είναι δυνατόν οι μεταρρυθμίσει για τι οποίε φέρουμε και εμεί κάποια ευθύνη. Αλλά εγώ είχα προειδοποιήσει δεν είναι δυνατόν να έχουμε περισσότερε στρεβλώσει του ανταγωνισμού από ό,τι είχαμε διαπιστώσει ποτέ στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιλέρα. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Για το πώς γίνονται οι άμεσες ενισχύσεις, πώς εφαρμόζεται το σύστημα άμεσων ενισχύσεων στα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, είδα τις, τους συγκριτικούς πίνακες, αρχίζουμε και βλέπουμε τα αποτελέσματα και στην Ισπανία. Από τους πίνακες ε, πάντως διαπιστώνουμε ότι κάθε κράτος, κάθε χώρα έκανε το δικό του κοστούμι, ανάλογα με τα μέτρα του, τις ιδιαιτερότητες της χώρας, τις προτεραιότητες κάθε κυβέρνησης. Έτσι διαμόρφωσε το σύστημα ώστε να το εξυπηρετεί. Το ο καθένας μπορεί να χαρακτηρίσει το σύστημα καλό, μέτριο, κακό. Πάντως συμφωνώ με τον κύριο Ντές ε, ότι έχουμε λιγότερο κοινή γεωργική πολιτική από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις. Ε, αμφισβητήθηκε πολύ το δικαίωμα ε, των ιστορικών κριτηρίων αναφοράς. Όταν εξετάζαμε τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, είπαμε ότι θέλουμε περισσότερη κοινωνική νομιμοποίηση των ενισχύσεων. Και για να δώσουμε τέτοια κοινωνική νομιμοποίηση δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο σε ιστορικά κριτήρια αναφορά στην ιστορική αντίληψη των καλλιεργιών. Γι' αυτό και προσθέσαμε ε, τις ενισχύσεις για τον greening, το πρασίνισμα της γεωργίας, τι ε, τις περιοχές οικολογικής εστίασης και διαπιστώσαμε από το τελικό αποτέλεσμα ότι και πάλι το κάθε κράτος έκοψε και έραψε στα μέτρα του το σύστημα. Δεν ξέρω αν η μεταρρυθμίση αυτή των άμεσων ενισχύσεων θα ε, επιφέρει την ε, απαραίτητη νομοποίηση ώστε να καταλάβει και να αντιληφθεί η κοινωνία ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τα γεωργικά εισοδήματα και τους Ευρωπαίους γεωργούς. Γιατί πραγματικά με πλήσει αυτή η διαφοροποίηση και η ποικιλομορφία, η πολυμορφία της εφαρμογής του συστήματος. Το μείζο πρόβλημα είναι το εξή. Ε, πώς θα εξασφαλίσουμε αξιοπρεπές χειρουργικό εισόδημα και κτηνοτροφικό εισόδημα. Νομίζω ότι χρειάζονται οι ενισχύσει. Εγώ είμαι υπέρ των άμεσων ενισχύσεων. Αλλά δεν θεωρώ ότι έχει εφαρμοστεί αποτελεσματικά το σύστημα. Ιδιαίτερα δεν ήταν θετική αλλαγή από τις ιστορικές αποδόσεις στο νέο σύστημα. Εγώ είχα περισσότερες προσδοκίες ε, για μεγαλύτερη νομοποίηση των νέων προτάσεων. Είχαν, δημιουργηθεί υψηλές προσδοκίες και, και για το θέμα του ενεργού Γιώργου, για το καθεστώς αυτό. Γιατί θέλουμε να στηρίξουμε τους γεωργούς που έχουν γεωργική δραστηριότητα, που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και πλούτο. Ίσως δεν υλοποιήθηκε απόλυτα αυτός ο στόχος, αλλά στην Ισπανία είπαμε να το σχετίσουμε αυτό το μέτρο με το εισόδημα. Βέβαια, το εισόδημα δεν μπορεί να είναι το αποκλειστικό κριτήριο για τις άμεσες ενισχύσεις. Αλλά η ύπαρξη δραστηριότητα στο αγρόκτημα, στο χωράφι, να είναι επαρκές κριτήριο για τη χορήγηση των άμεσων ενισχύσεων. Οπότε θα πρέπει ε, νομίζω ότι χάσαμε το παιχνίδι σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση αυτής της μορφής του ενεργού γεωργού για να αυξήσουμε την ε, νομιμοποίηση των άμεσων ενισχύσεων. Νομίζω ότι είναι σφαλμένη η πρόταση της ε, Ισπανικής κυβέρνησης να συνδεθεί η ιδέα του ενεργού γεωργού με το εισόδημά του αποκλειστικά και μόνο ποιο θα πρέπει να είναι το γεωργικό εισόδημα ενός γεωργού για να δικαιούται περισσότερη ή λιγότερη ενίσχυση. Επίσης, περιφερειοποίηση. Στην Ισπανία ίσχυσε η περιφερειοποίηση. Αλλά εσείς ε, πολλαπλασιάσατε, διπλασιάσατε την πρόταση της Ισπανικής κυβέρνησης. Μέχρι και 50 περιφέρειες ε, προτείνατε. Κάτι που δημιουργεί ανασφάλεια στους γεωργούς. Μέχρι τον Οκτώβριο πρέπει να περιμένουν και πάλι δεν θα γνωρίζουν με ακρίβεια πώ θα δοθούν οι άμεσες ενισχύσει. Πολλές αβεβαιότητες δημιουργούνται με την παρούσα κατάσταση. Και τέλος, ε, λυπούμε πολύ, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στο σύστημα των άμεσων ενισχύσεων, αλλά με τη μεταρρύθμιση αυτή δεν επιτύχαμε ούτε την νομιμοποίησή τους, ούτε την διασφάλιση των ε, γεωργών που έχουν τη γεωργική δραστηριότητα ως κύρια απασχόληση ε, και την παραμονή τους στην Ήπεθρο. Προσοχή, γιατί αυτό το κόψιμο και ράψιμο που έκανε το κάθε κράτος με, τις ανάγκες, με βάση τις ανάγκες του, δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα φέρει στην ενιαία μας αγορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Χόισλινγκ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Νομίζω ότι το ότι έχουμε διαφορετικά μέτρα σε διάφορα κράτη-μέλη είναι αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου. Βεβαίως λοιπόν αγαπητέ έχουμε και εμείς ένα τμήμα της ευθύνης, είμαστε συνομοθέτες. Εάν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προτείνουν προσαρμογές ταχύτερες στο δικό μας επίπεδο στα νέα κράτη-μέλη, από ό,τι εμείς επιτύχαμε στα παλιά κράτη-μέλη, τότε φέρουμε κι εμείς την ευθύνη. Και το ότι υπάρχουν τόσε εξαιρεσει σε μεγάλο βαθμό είναι ευθύνη των κρατών μελών διότι θέλησαν να εφαρμόσουν με τη δική τους προσέγγιση το πρασίνισμα. Τώρα έχει έννοια αυτό. Ή η Κομισιόν θα πρέπει να δει τι έννοια ακριβώς έχει αυτό το greening. Όμως δεν θα συμπέρανα ότι η ΚΚΠ είναι τώρα πιο άνηση από ό,τι προηγουμένως. Θα έλεγα ότι οδεύουμε προς μία ομογενοποίηση. Περιορίσαμε τη χρήση των στοιχείων του παρελθόντος. Εάν κάποιος παλιά είχε κάποια απέτηση πληρωμής, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να την έχει ΕΣΑΗ θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει αυτές τις προσαρμογές βέβαια ταχύτερα, αλλά νομίζω ότι η προσέγγιση των ε, ενισχύσεων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κάτι περίπλοκο. Γενικά λοιπόν δεν θα συμφωνούσα ότι οι προτάσεις αυτές οδηγούν σε περισσότερες αποκλίσεις μεταξύ της Ευρώπης. Πιστεύω ότι είναι λυπηρό ότι δεν θα έχουμε το 2020 το ίδιο σύστημα, αλλά το 2020 θα έχουμε όλοι αναλάβει την υποχρέωση να κάνουμε μια νέα μεταρρύθμιση. Θα δούμε αν μπορούμε να επιτύχουμε αυτήν την ομοιομορφία. Και βεβαίως πάντα θα υπάρχουν και επιμέρους ε, απαιτήσει για διαφοροποιήσεις και αυτό θα δημιουργεί δυσχέρειες θα πρέπει όμως να ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε να επιτύχουμε. Θέλουμε σε κάθε κράτος μέλος να υπάρχει η ίδια ακριβώς προσέγγιση. Αγαπητέ συνάδελφε Ντες, και στη Γερμανία έχουμε 16 διαφορετικές πρακτικές ε, εφαρμογής. Στη Βαβαρία εφαρμόζουν αλλιώς το δεύτερο πυλώνα από ό,τι στο Σλέσφι Χόλσταϊν. Αυτό είναι θέμα ευθύνη ε, των περιφερειών και δεν νομίζω ότι είναι κατά Δεν ήθελα να σας περιορίσω, αλλά εφαρμόστε μόνοι σας κάποια αυτοπιθαρχία στη χρήση του χρόνου. Ο κύριος Γιάρ. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Σωστό. Ε, συμμετείχαμε στην απόφαση αυτού του νομοθετήματος. Και υπόθηκε ότι υπάρχουν πολλές διαφορές Και βεβαίω τα κράτη-μέλη αξιοποίησαν κάθε δυνατότητα με πολύ καινοτόμο τρόπο. Και βεβαίω κατά τη γνώμη μου έχει αυξηθεί η διαφορετικότητα. Και θα πρέπει όταν θα κάνουμε την επόμενη μεταρρύθμιση να δούμε αν θέλουμε μια κοινή γεωργική πολιτική. Για τελειώ να καταργήσουμε το κοινή. Και ένα ερώτημα που έθεσαν και άλλοι συνάδελφοι. Εάν είναι τόσο διαφορετικέ οι γεωργικέ πολιτικέ, γιατί πρέπει να στέλνουμε τα χρήματα στι Βρυξέλλε για να τα μοιράζουν. Και κάτι άλλο. Είμαι αντίθετο, κύριε Χόισλινγκ. Βεβαίω πάντα υπάρχει αυτή η αντίθεση κοινή πολιτική, περιφερειακές διαφορές. Αλλά η κοινή στρατηγική είναι ο πρώτος πυλώνας, το πρασίνισμα. Όταν ήμουν νέος ε, πρόσφατος ε, κοινοβουλευτικό έτσι κατάλαβα την κοινή γεωρική πολιτική. Ο πρώτος πυλώνας είναι το κοινό στοιχείο που δεν πρέπει να κλονιστεί. Αυτό πρέπει να είναι η κοινή χρηματοδότηση και πρέπει να είναι 100% η κοινοτική χρηματοδότηση. Και μετά έχουμε το δεύτερο πυλώνα για να λάβουμε υπόψη τι περιφερειακέ διαφορέ, αλλά εκεί πρέπει να υπάρχει συγχρηματοδότηση, γιατί είναι χρηματοδότηση ε, που έχει να κάνει με τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Αλλά με το πρασίνισμα δεν είναι σαφής αυτή η διαφοροποίηση. Εγώ λυπάμαι για τη σημερινή κατάσταση. Παρόλα αυτά δέχομαι και την ευθύνη μου. Θα πρέπει λοιπόν να κάτσουμε μαζί για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και μια τελευταία ερώτηση στην Κομισιόν. Θεωρείτε ότι έγινε, έγινε πιο πολυπίκυλη η γεωρική πολιτική ή έχει γίνει πολύ πιο άχρωμη. Πείτε μας ποια είναι η εντύπωσή σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούντα. ο Μπούντα. Uh, ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ για την παρουσίαση από πλευρά τη Επιτροπή. Εκτιμώ την θέση της ότι πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις των κρατών μελών για τις απευθείες ε, ενισχύσεις, για τις άμεσες ενισχύσεις. Ωστόσο θα πρέπει να παρεμβαίνει η Επιτροπή όταν διαπιστώνει παρεκκλήσεις κάποιων κρατών μελών. Θα ήθελα όλα να γίνουν καλά στη χώρα. Δεν θέλω να πάει κακά η κατάσταση, αλλά σε ό,τι αφορά την χειροτροφία και τα πουλερικά, η κυβέρνηση δεν ζήτησε πόρους για την ευημερία των ζώων εδώ και πολλά χρόνια. Κινδυνεύει να χάσει τα χρήματα για πάντα, διότι σε άλλα κράτη-μέλη η ευημερία των ζώων χρηματοδοτείται περισσότερο. Επίσης θα έπρεπε στο μέλλον να υπάρξει σχέση μεταξύ πραγματικής παραγωγής και άμεσων ενισχύσεων. Δηλαδή, μια ομάδα γεωργών της χώρας μου ήθελε να εισάγει δεν ενδιαφέρει από ποια χώρα, κάποια ζώα. Ωστόσο, δεν βρήκε ζώα που κάλυπταν τα κριτήρια που ήθελε, γιατί στη χώρα εκείνη υπήρχε μικρό ενδιαφέρον για την ευημερία των ζώων. Αυτό είναι ο λόγος τον οποίο πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της, των άνεμων ενισχύσεων και της πραγματικής παραγωγής. Ευχαριστώ. Δεν είναι η στιγμή να κάνουμε απολογισμούς. Η μελέτη είναι προφανώ πολύ ενδιαφέρουσα. Την ευχαριστώ την Επιτροπή και τον κύριο Πασκού που δυστυχώς μας οδηγεί στο να διαπιστώσουμε αυτό που φοβόμασταν εν μέρη. Ότι υπάρχει δηλαδή μια χρήση από πλευράς των κατώμερων της ευελιξίας για να αποφύγουν περισσότερο τον επί τον ε, ε, αντίκτυπο των ε, αλλαγών. Δηλαδή χρησιμοποιήθηκε η ευελιξία για να δημιουργηθεί αυτό το διαφοροποιημένο με μοσαϊκό που δημιουργήσε μια σειρά προβλημάτων, μια μικρότερη κοινή πολιτική ή μεγαλύτερες διαφορές ανάμεσα στα κράτη. Εμείς έχουμε την ευθύνη εν πολλής, διότι η μεταρρύθμιση για πρώτη φορά έγινε με συνεισφορά και του Κοινοβουλίου. Εμείς ζητούσαμε μεγαλύτερη ευελιξία στους τριμερείς διαλόγους για να αποφύγουμε να πάμε σε μια κατεύθυνση που δεν θέλαμε. Δημιουργήθηκε λοιπόν αυτός ο φαύλος κύκλος. Τι να κάνουμε. Το ερώτημά μου είναι τι κάνουμε τους επόμενους μήνες με την εφαρμογή τα κράτη-μέλη σίγουρο είναι θα προσπαθήσουν να επανέλθουν στην προσαρμογή περαιτέρω προσαρμογή της πρακτικής εφαρμογής ε, των πολιτικών και θα πούν μειώνουμε το συνδεδεμένο τμήμα, αυξάνουμε το υποχρεωτικό τμήμα. Όλα αυτά δεν δημιουργούν τον κίνδυνο να φέρουν ακόμα μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις στην εφαρμογή της ΚΑΠ. Είναι, χρειάζεται νομίζω στη φάση αυτή να κάνουμε μια ενδιάμεση επανεξέταση της κατάστασης. Να δούμε, έγιναν λάθη. Μπορούμε να τα διορθώσουμε. Ευχαριστώ. Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με προσοχή και ιδιαίτερα ενδιαφέρον την παρουσίαση και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την ενημέρωση. Η νέα περίοδος ε, του συστήματος άμεσων ενισχύσεων έχει ξεκινήσει και από τη στιγμή που λάβουν τις αποφάσεις τα κράτη-μέλη θα ενημερωθούν και οι πολίτες. Φυσικά υπάρχουν μερικές διαφορές, μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και βλέπουμε ε, σε μερικούς πίνακες 5-6 διαφορετικές ομάδες και δύσκολο είναι να προβλέψουμε από τώρα ποια κράτη-μέλη θα έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα ή τα χειρότερα. Κοιτάζοντας και από τη χώρα μου, ε, διαπιστώνω ότι μερικές χώρες ε, θα καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες να προσαρμοστούν σε νέο μηχανισμό, ενώ άλλες χώρες θα κάνουν όσο λιγότερες αλλαγές μπορούν, εφαρμόζοντας μια πιο αμυντική συμπεριφορά. Ρωτώ λοιπόν, ποιες χώρες ε, ήταν ε, πιο αποτελεσματικές και επιτυχείς ε, στην εισαγωγή του κανονισμού και ποιες προτίμησαν να παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό στο παλιό σύστημα. Ξέρω ότι η Ρουμανία άψε την αξιολόγηση του πρασινίσματος και στήριξε ε, τις μεσαίες περισσότερο ε, εκμεταλλεύσεις, των 30 εκταρίων. Αυτό ήταν ο κοινό παρανομαστής. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τη βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων, ε, μια και εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο το σύστημα άμεσων ενισχύσεων στα κράτη-μέλη. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήδη υπόθηκε ότι είχαμε την κοινωνικοποίηση του συστήματος μετά την οικολο... οικολογοποίηση του συστήματος αλλά γι' αυτό μήπως δεν έχουμε τόσο πολύ εθνικό περιθώριο δράσης επειδή ακριβώς δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε σε μια πιο οικολογική, πιο κοινωνική γεωρική πολιτική. Τώρα, αν αυτά τα περιθώρια εθνικών ε, ελιγμών είναι καλά ή άσχημα, δεν θέλω να κρίνω. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης. Πρώτα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί και μετά θα έπρεπε να κάνουμε μια έντιμη ενδιάμεση αποτίμηση να δούμε τι θα έχει λειτουργήσει, τι θα έχει επιδράσει, εάν ό,τι έχει επιτευχθεί είναι σύμφωνο με τους στόχους ε, της κοινή γεωρικής πολιτικής και σε τι βαθμό όχι. Μόνο αν έχουμε αυτή τη σωστή αποτίμηση μπορούμε να καθορίσουμε σωστά την επόμενη κοινή γεωρική μας πολιτική για μετά το 20. Θα πρέπει μετά να επανακαθορίσουμε τι γεωργία θέλουμε τι θέλουμε να επιτύχει η γεωρική μας πολιτική, τι θέλουμε να επιτύχουμε πέρα από την προώθηση, της, την ενίσχυση των εκμεταλλεύσεων, δηλαδή διατήρηση της υπαίθρου, οικολογικές πολιτικές κτλ. Και τότε μόνο μπορούμε να καθορίσουμε νέες καθευθυντήριες γραμμές. Είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστούμε το χρόνο αν ε, ζητάτε το λόγο τελευταία στιγμή αφού έχουμε κλείσει τον κατάλογο. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δυστυχώς απουσίαζε από το πρώτο τμήμα της παρουσίασης. Αλλά νομίζω ότι δίκαιο έχει ο Παόλο Δεκάστρο ότι και εμείς ε, υπερψηφίσαμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις ε, δεν θα πρέπει να ανύπτουμε τώρα τα σχήρα μας για τα αποτελέσματα. Ήταν πολύ χρήσιμη παρουσίαση για την κατάσταση ε, και είναι πρόωρο να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της των μεταρρυθμίσεων. Το θέμα είναι το greening θα ε, λειτουργήσει και αν δεν αποφέρει ε, τις περιβαλλοντικές συνέπειες που ζητούμε, τι θα γίνει, ποιες θα είναι οι συνέπειες. Μπορούμε και στο greening, στο πρασίνισμα να εφαρμόσουμε κάποια απλούστευση. Και μία διευκρίνηση θα ήθελα να κάνετε πόσες ε, από τις 28 χώρες θα έχουν ε, ομοιόμορφο σύστημα πληρωμής ανεκτάριο μέχρι ε, είτε με είτε περιφερειακές πληρωμές είτε σε βάση καλλιέργειας. Ήθελα αυτή την ερώτηση να μου απαντήσετε. Κύριος Μπόγκοβιτς. Ευχαριστώ πρόεδρε πολύ καλή η έκθεση. Στο μέλλον θα έπρεπε να έχουμε πιο συγκεκριμένες εικόνες για το πώς λειτουργεί το σύστημα. Επίσης θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι συμβαίνει όταν μετά από αυτό που μας είπε ο καθηγητής πριν τη σύγκριση για την, ε, μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωση. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα γενική συζήτηση για το θέμα αυτό, TTIP, διαχείριση κινδύνου, εν ώψη των ε, επερχόμενων συμφωνιών Ένωσης και ΙΠΑ και των αλλαγών που αυτές θα φέρουν στην γεωργία, γίνεται όλο και πιο εμφανές το πόσο διαφοροποιημένες είναι οι πολιτικές και πόσο δύσκολο είναι για τους δικούς μας γεωργούς να ανταγωνιστούν τους Αμερικανούς γεωργούς και τις ανταγωνιστικές και επιθετικές τους πολιτικές από την οπτική γωνία της αμυντικής στάσης που αυτή τη στιγμή έχουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντρίε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πασκό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωση. Φάνηκε ότι ε, μερικές φορές χρησιμοποιούμε τα μέσα αλλά άσχετα με τους κοινούς μας στόχους. Και το θέμα δεν είναι το σύνολο των μέσων που τα εγκρίναμε υπερψηφίζοντας τη μεταρρύθμιση. Το θέμα είναι αν έχουμε θέσει τι σωστέ ερωτήσει ε, για τους ε, κοινούς στόχους και αν είμαστε σε θέση σήμερα να έχουμε ένα κοινό στόχο της κοινή γεωργικής μας πολιτικής. Αυτό μας ε, ενδιαφέρει κατά την εφαρμογή του, του οικονομικού ή του γεωπονικού μοντέλου, που δεν είναι ενιαίο. Δεν ξέρω αν είχαμε αρκετά καλή προετοιμασία ώστε να ξέρουμε προς τα αποβαδίζουμε. Και αυτό είναι ένα θέμα που επανέρχεται. Στα πλαίσια της μελλοντική μεταρρύθμισης ε, θα πρέπει κατά προτεραιότητα αυτό να βρούμε. Να μην περιμένουμε τις ενδιάμενες αξιολογήσεις για να προβληματιστούμε για το τι είδους γεωργία θέλουμε σήμερα και τι γεωργία θέλουμε για το μέλλον. Ποιον θέλουμε να ωφελήσει η γεωργία, για ποιο λόγο και η περαιτέρω πορεία θα, θα εξαρτηθεί από την απάντηση αυτών των ερωτημάτων. Αυτέ τι βασικέ ερωτήσει που έχουν διαρθρωτική σημασία θα πρέπει πρώτα να απαντήσουμε, γιατί θα διαμορφώσουν την κοινή γεωρική πολιτική. Άσχετα με τη, τη μηχανική, το σύστημα που θα εφαρμόσουμε και τα μέσα. Πρώτα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τα όρια που έχει αυτή η διαδικασία στην οποία συμμετείχαμε και να δούμε και ποιες προοπτικές έχει. Αυτά είναι μείζωνα πολιτικά θέματα για το ποιο είναι ο κοινό μα στόχος και πώς θα τον εφαρμόσουμε προς ε, όφελος ε, των γεωργών μας και των περιφερειών μας. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ να πω δύο λόγια. Η γεωργία μας χαρακτηρίζεται από τεράστια πολυμορφία. Άλλη γεωργία του Νότου, άλλη γεωργία του Βορρά, άλλη γεωργία στις παλιές χώρες μέλη, άλλη στις καινούριες. Έχουμε μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μικρές. Τεράστια διαφορά, τεράστια πολυμορφία γι' αυτό και θέλουμε ελαστικότητα. Έχουμε διάφορες ψηφίδες σε ένα τεράστιο ψηφιδωτό. Γι' αυτό και ζητούμε ελαστικότητα. Μα είπατε ότι κάθε χώρα ε, ε, ράβει το κουστούμι στα μέτρα του. Το θέμα είναι τι υλικό θα επιλέξουμε για αυτό το κουστούμι και το υλικό και ο τρόπος με τον οποίο ράβουμε το κουστούμι το αποφασίσαμε όλοι από κοινού. Υπάρχει και το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Την εξασφαλίζουμε, όχι ακόμη. Θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη όμως και εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα των γεωργών μας. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα στρέμμα με ελαιόλαδα, ε, με, με ελαιόδεντρα, συγγνώμη, με ένα στρέμμα με δημητριακά ή ένα στρέμμα χορτονομής. Θα πρέπει λοιπόν ε, να, αναλύσουμε αυτή την κατάσταση και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Σίγουρα θα μπορούσαμε να θετήσουμε και διαφορετική λύση. Θα ήταν όμως καλύτερη, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Γιατί τώρα ε, προβαίνουμε σε αυτή την πρώτη αξιολόγηση. Και σίγουρα θα πρέπει να ζητήσουμε το πρασίνισμα, τη φιλοπεριβαλλοντική γεωργία και να τη διευκρινίσουμε, γιατί υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες εδώ και αμφισημίες και προβληματίζονται οι γεωργοί, δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Επίσης, έχουμε, εξακολουθούμε να έχουμε κοινή αγροτική πολιτική. Ε, θα πρέπει να είναι πιο ομοιόμορφη ή καλό θα είναι να είναι διαφοροποιημένη. Και ας μην λέμε συνέχεια ότι δεν έχουμε κοινή γεωρική πολιτική. Γιατί έχουμε και νομίζω ότι είναι πιο δίκαια. Απλώς έχουμε διοικητικά προβλήματα και υπερβολικές διοικητικές διατυπώσεις για το πρασίνισμα. Τώρα, αν είναι καλύτερο το σύστημα, θα το δείξει ο χρόνος. Αυτά και ευχαριστώ τον ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον οποίο και ξαναδίνω το λόγο για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο. Ευχαριστώ για όλες τις παρεμβάσεις σας, τα σχόλια και τις ερωτήσεις που τέθηκαν, για τη συζήτηση ιδίως που έγινε, την αντιπαραβολή διαφορετικότητας και κοινών πολιτικών. Καταρχάς να σας πω ότι αυτό που παρουσιάσαμε σήμερα αντικατοπτρίζει τις αποφάσεις πολιτικής που έλαβαν τα κράτη-μέλη για το πώς θέλουν να εφαρμόσουν το νέο σύστημα άμεσων ενισχύσεων. Σε δύο-τρία χρόνια θα δούμε το αποτέλεσμα της πολιτικής και πόσο συγκεκριμένα συμφώνησαν οι παραγωγοί να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Είναι νομίζω πρόημο να κρίνουμε αυτή τη στιγμή την επίδοση του συστήματος. Η είναι αναμενόμενη ωστόσο αυτή η διαφορετικότητα και το είπαν πολλά μέλη της Επιτροπής μετά από αφού υιοθετήθηκαν νέοι στόχοι πολιτικής που όπως είδαμε συνοδεύονταν από μια βούληση να έχουν μια πιο αποτελεσματική πολιτική που θα αντικατοπτρίζει διαφορετική, τη διαφορετική κατάσταση της γεωργίας. Παραγωγή, ανταγωνιστικότητα, επίπεδο υποστήρι, κρατικής υποστήριξης, τύπο κρατικής υποστήριξης. Όλα αυτά εξαρτώνται από την τοπική περιφερειακή κατάσταση. Είναι σαφές, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε τη διαφορετικότητα αυτή και να την διατηρήσουμε μέσω ενός περιορισμένου κανονιστικού πλαισίου αυτό που έχουμε, ε, περιορισμένων δημοσιονομικών δυνατοτήτων, αυτό έχουμε, και το να εξετάσουμε πώς θα εφαρμόσουμε αυτή τη νέα πολιτική. Ωστόσο η πρόκληση για τους γεωργούς και ο στόχος της πολιτικής για την ασφάλεια και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, αλλά και την συνεισφορά στην εδαφική ισορροπία, η στόχη αυτή είναι κοινή. Το θέμα είναι πώς τα κοινά εργαλεία θα τα εφαρμόσουμε για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, αλλά πρέπει να τα, να τα προσαρμόσουμε και εδώ είναι η ευελιξία που έχουν τα κράτη-μέλη, να τα προσαρμόζουν στη συγκεκριμένη κατάσταση για να πετύχουν αυτούς τους ε, στόχους πολιτικής. Δύο λόγια τώρα για την ε, διαφορετικότητα. Αυτή η διαφορετικότητα δεν σημαίνει περίπλοκα συστήματα. Υπάρχουν μια σειρά επιλογών για το greening, για παράδειγμα, αλλά δεν νομίζω ότι ε, αμελούμε την απλοποίηση. Απλά τα κράτη-μέλη πρέπει να βρουν μια ισορροπία μεταξύ σωστής διαχείρισης και απλών διαδικασιών. Η διοίκηση χρειάζεται απλές διαδικασίες, το ίδιο χρειάζονται και οι γεωργοί. Δύο λόγια για την παρέμβαση, την εμπλοκή της Κομισιόν στις αποφάσεις των κρατών μελών. Θα ήθελα να πω, το είπα, ότι η Κομισιόν δεν έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίπτει αποφάσεις των ε, κρατών μελών. Τους τελευταίους μήνες βοηθά, υποστηρίζει τα κράτη-μέλη... στις προσπάθειές τους να μεταφέρουν στην ουσία τις επιλογές πολιτικής ένα σύστημα εθνικό που συμφωνεί με το κανονιστικό πλαίσιο. Γι' αυτό έχουμε και όλες αυτές τις ε, διαφοροποίησεις. Αλλά οι επιλογές που έκαναν τα κράτη-μέλη για την εθελούσια ε, υποστήριξη για τους, ε, γεωργού, την, την, υποστήριξη των γεωργών σχετίζονται όλα με τις επιλογές πολιτικής. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να περιγράψουμε και που είμαστε σε, λίγα, σε λίγες αυτές διαφάνειες είναι πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση και πόσο διαφορετική είναι ε, η θέση του γεωργού από κράτος σε κράτος. Πρέπει η πολιτική να έχει κάποιες ε, εγγυήσεις αλλά ταυτόχρονα κάποιες, ε, ε κάποιες τροχοπέδες μια τελευταία παρατήρηση. Αυτό που είπε η Ισπανίδα συναδελφός για τους ενεργούς γεωργούς. Αυτό είναι προβληματικό θέμα. Το άρθρο 9 του βασικού κανονισμού δεν πληρεί τους στόχους πολιτικής πλήρως να δίνει έμφαση στο ότι απευθείας ενισχύσεις παίρνουν, άμεσες ενισχύσεις παίρνουν οι γεωργοί που παράγουν που κάνουν δραστηριότητε που σχετίζονται με την διατήρηση της γης σε μια καλή κατάσταση περιβαλλοντική και για να μπορέσει να παράγει. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε λοιπόν την σύνδεση των άμεσων ενισχύσεων με το επίπεδο που, των εισοδημάτων που δημιουργούνται από τη γεωργία. Τώρα, αν υπάρχουν καλά ή κακά κράτη-μέλη, δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό εξαρτάται από τους πολιτικούς στόχους που έχει κάθε κράτος και που σχετίζονται με την επιλογή πολιτικής. Δεν θα έρθει η Κομισιόν να κάνει αν η δημόσια υποστήριξη που διαμορφώθηκε σε το επίπεδο είναι καλή ή όχι. Και θα σταματήσω εδώ. Także e, proszę Σίγουρα θα πρέπει να συνεχίσουμε την παρακολούθηση, την ανάλυση και παρακαλούμε να μας ενημερώνετε τακτικά για τον τρόπο εφαρμογής του συστήματος άμεσων ενισχύσεων. Περνάμε στο επόμενο σημείο και πάλι παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκβασης των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου για την αμοιβαία προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Θα δώσουμε το λόγο στην ε, αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη, την κυρία Μονίκ Παριά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ κάθομαι και εδώ θα παραμείνω. Αν μου επιτρέπετε για να μην αλλάζουμε θέση και χάνω χρόνο. Σήμερα το πρωί στις συζητήσεις ε, που έγιναν για τη διατλαντική εταιρική σχέση, πολλοί μιλήσατε για τη σημασία που έχουν οι γεωγραφικές ενδείξεις. Και με ιδιαίτερη χαρά θα σας δώσω μια εικόνα και μια επισκόπηση της έκβασης των διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Μαρόκου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Η συζήτηση αυτή μονογράφηκε στις 6 Ιανουαρίου στο Βερολίνο στα πλαίσια της έκθεσης ε, για τη Γεωργία στην Πράσινη Εβδομάδα παρουσία του Πρόεδρου του Επιτρόπου Χόγκαν και του Υπουργού Γεωργίας του Μαρόκου Ακανούς. Ε, η συμφωνία εντάσσεται στην εντολή που έδωσε το Συμβούλιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2005 για την ευάθυνση στις γεωργικές ε, δοσμολογικές παραχωρήσεις. Οι διαπραγματεύσεις σε μια πρώτη φάση αναφέρθηκα στην απελευθέρωση των ε, γεωργικών προϊόντων και μετά την ε, διεκπαιρέωση αυτών των διαπραγματεύσεων και μετά την θέση εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2012 της Γεωργικής Συμφωνίας ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Το Δεκέμβριο του 2012 συγκεκριμένα. Ένα άρθρο της ε, Γεωργικής Συμφωνίας προέβλεπε την έναρξη των διαπραγματεύσεων ε, ε, μέσα στο τρίμηνο που ακολουθεί, της, ε, θέση ισχύ, ακολουθεί τη θέση ισχύ της συμφωνίας. Έγιναν πολύ κύριοι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Δεκεμβρίου του 2012 και του Νοεμβρίου του 2014. Και οι πιο ουσιαστικέ συζητήσει έγιναν μεταξύ Δεκεμβρίου 2012 και Φεβρουαρίου 2014. Και Έκτοτε και μέχρι το τέλος του 2014 είχαμε μία παύση. Εκεί είχαμε κάποιες διαφορές με το Μαρόκο σε ό,τι αφορά τις κανονιστικές μεταρρυθμίσεις που χρεια... ήταν απαραίτητες για τους τρόπους εκτελονισμού των απορροκυπευτικών. Ιδιαίτερα για τις δομάτες ε, που ε, υπόκεινται σε τιμή εισόδου χρειάστηκαν κάποιες τεχνικές λύσεις για τις διαδικασίες εκτελονισμού και την ε, καταποκοπή αξία της εισαγωγής. Τελικά το Μαρόκο συμφώνησε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις ε, για τις γεωγραφικές ενδείξεις και χρειάστηκε ελάχιστο χρόνο ε, για να διεκπαιρεώσουμε αυτέ τι συζητήσει και να καταλήξουμε σε μια πολύ ικανοποιητική συμφωνία, ιδιαίτερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί χάρη στη συμφωνία αυτή θα εξασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας ε, για 3.200 ε, ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις στο Μαρόκο και 30 μαροκινές γεωγραφικές ενδείξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 14 γεωγραφικές ενδείξεις για τρόφιμα και 16 για κρασιά. Πρόκειται για μια κλασική συμφωνία γεωγραφικών ενδείξεων με την ίδια δομή που είχαν οι πρόσφατες συμφωνίες που συνάψαμε με τη Γεωργία και τη Μολδαβία. Εξασφαλίζει άμεση προστασία όλων των γεωγραφικών ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας στο Μαρόκο, χωρίς μεταβατική περίοδο και επιτρέπει η συμφωνία αυτή άμεση προστασία. Δεν χρειάζεται μεμονωμένη η ατομική καταγραφή των γεωγραφικών ενδείξεων για να ενεργοποιηθεί αυτή η προστασία. Το Μαρόκο φυσικά μπορεί να εφαρμόσει τις εσωτερικές του διαδικασίες για την ε, καταγραφή αυτών των ενδείξεων, αλλά δέχτηκε αλλά ε, συμφώνησε να δεχτεί αυτή την καταγραφή χωρίς επιπλέον διοικητικές δαπάνες ε, για την Ευρώπη προβλέφθηκε μάλιστα και τακτική ενημέρωση των παραρτημάτων ε, για να προσθεθούν νέε γεωγραφικές ενδείξεις χάρη στην επικαιροποίηση και μάλιστα ο κατάλογος που περιλαμβάνεται στο σχέδιο συμφωνίας είναι ο κατάλογος που οριστικοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου του 2013. Στο μεταξύ όμως προέκυψαν και νέες γεωγραφικές ενδείξεις που δεν υπάρχουν προς το παρόν στον κατάλογο αλλά θα περιληφθούν ε, στην πρώτη συζήτηση της Μικτής Επιτροπής ε, που είναι επιφορτισμένη με την επικαιροποίηση του παραρτήματος. Ε, έχει επισυναφθεί στη συμφωνία αυτή και μια κοινή δήλωση που περιλαμβάνει μια σειρά δεσμεύσεων των δύο συμβαλωμένων μερών. Για παράδειγμα, να μην ζητηθούν τέλη καταγραφής των γεωγραφικών ενδείξεων. Επίσης, προβλέπεται τεχνική παρακολούθηση ε, στο Μαρόκο για την προώθηση και την ανάπτυξη των γεωγραφικών ενδείξεων στην Μαροκινή Επικράτεια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια προγράμματα διαφήμισης, προβολής και προώθησης και επίσης ένα σημαντικό θέμα, ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των συμβαλωμένων μερών. Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που αφορούν τις ονομασίες προέλευσης ή τι γεωγραφικές ενδείξεις στα πλαίσια της Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου ή στα πλαίσια της Συμφωνίας της Λισαβόνας της Παγκόσμια Οργάνωσης Πνευματική Ιδιοκτησία. Ε, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τη συμφωνία αυτή γιατί ενισχύει τη, τα ποιοτικά γεωρικά προϊόντα και τις εξαγωγές μας και επίσης ανοίγει το δρόμο για άλλες παρόμοιες ε, συμφωνίες με την Αλγερία, την Τινησία, το Λίβανο, με άλλες χώρες δηλαδή της περιοχής και μάλιστα δημιουργεί ένα θαυμάσιο προηγούμενο η συμφωνία αυτή για την προσέγγιση που θέλουμε να προωθήσουμε και να ενισχύσουμε σε ό,τι αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και την ε, αναβάθμιση και αξιοποίησή τους. Επίσης ενισχύει τις εμπορικές μας σχέσεις με το Μαρόκο, που πέρυσι είχαν κάπως δεινοπαθήσει εξαιτία του προβλήματος που είχαμε με τις ντομάτες. Δύο λόγια για τα διαδικαστικά. Εκπονούμε δύο σχέδια απόφασης, το ένα για την υπογραφή και το δεύτερο για την ε, σύναψη της συμφωνίας, την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Έχετε λάβει αυτά τα δύο σχέδια απόφασης θα πρέπει ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την απόφαση για την ολοκλήρωση για την ε, σύναψη της συμφωνίας στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Διευθύντρια. Παρακαλώ, ποιος θέλει το λόγο για ερωτήσεις. Το θέμα είναι σημαντικό, δύσκολο, αλλά τελικά φαίνεται ότι φέραμε σε αίσιο πέρα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και μάλιστα είναι υποδειγματική αυτή η συμφωνία και θα γίνει και πρότυπο για παρόμοιες ε, συμφωνίες και με άλλες χώρες. Μιλήσαμε το πρωί για το TTIP. Τώρα έχουμε το Μαρόκο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο για σύντομα σχόλια στην κυρία Αγγιλέρα, μετά στην κυρία Σένερα και ούτω καθεξής. Κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσει προς την εκπρόσωπο τη Επιτροπή, ευχαριστώντας την για την παρέμβαση και τις πληροφορίες που μα έδωσε. Η συμφωνία με το Μαρόκο πρέπει να το δούμε θετικά, αλλά για την Ανταλουσία, την περιφέρειά μου, δεν είναι και πολύ θετικό. Γιατί προφανώς έχουμε ανταγωνιστικές παραγωγές. Αν έχετε τα στοιχεία παρακαλώ να μου τα δώσετε. Ήθελα το εξή. Ποιε είναι, εσείς μιλήσετε για συμφωνίες σχετικά με τις μεθόδους υπολογισμού της αξίας της τιμής της ντομάτας. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η τιμή της αξίας εισόδου της ντομάτας που έχετε συμφωνήσει με το Μαρόκο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε ακριβώς. Αν δεν το ξέρετε τώρα, κανένα πρόβλημα. Οι πληροφορίες που έχω εγώ ανέβηκε με διάφορες ε, παραγωγές ε, ποικιλιών ντομάτα, στην ντομάτα τσέρι για παράδειγμα. Οι παραγωγοί θέλουν να ξέρουν τα συγκεκριμένα στοιχεία, δεν ξέρουν ποια είναι η τιμή εισόδου αυτή τη στιγμή με τη νέα συμφωνία με το Μαρόκο. Για την ντομάτα λέω. Αυτό το προϊόν συγκεκριμένο. Δεύτερον, Είπατε ότι η συμφωνία μπήκε για τις γεωργιακές ενδείξεις και ονομασίες θα εγκρίθηκαν στις 9 Ιανουαρίου του 2013. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Δύο χρόνια δηλαδή. Αυτά τα δύο χρόνια δεν είναι και πολύ ενημερωμένος ο κατάλογος αυτό δημιουργεί κάποιες ζημίες, κάποια προβλήματα. Πέρασε δύο χρόνια για να οριστεί κάποια ονομασία. Καταλαβαίνω ότι λόγω της διάρκειας της, ε, των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ε, πάντα μένει κάτι απ' έξω. Αλλά είπατε εσείς ότι δύο χρόνια έγιναν οι συζητήσει αυτό το τελευταίο έτο ότι είχε αναγνωριστεί δεν θα μπει στον κατάλογο αυτό. Δεν έχει μπει στο κατάλογο αυτό. Πώ θα το λύσετε αυτό, Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η πρώτη σα ερώτηση ήταν εκτό θέματο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το κρίνει η διευθύντρια. Η κυρία Σένερ έχει τώρα το λόγο. Eh, eh. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Κοιτάξτε, κάθε φορά που έρχεται η Κομισιόν να μας εξηγήσει τι διαπραγματεύσεις κάνουν, τι εμπορικές συμφωνίες διαπραγματεύονται, δεν μας εξηγούν αρκετά. Θα ήθελα να μάθω τα εξής δύο. Πρώτον, όπως είπε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, φαίνεται ότι έχουμε προχωρήσει ε, επειδή υποχωρήσαμε στο θέμα της ντομάτας. Θέλω να σας πω ότι στη χώρα μου, στη Γαλλικία, παράγουμε και ντομάτες και άλλα χορταρικά και αισθανόμεθα τις επιπτώσεις της συνεχούς πτώσης της τιμής της ντομάτας. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε πώς προστατεύουμε την ε, ονομασία προέλευσης. Δεν καταλαβαίνω πώς διαπραγματεύεστε και πώς προστατεύετε τις ονομασίες προέλευσης. Τι θα κάνετε θετικό ή αρνητικό για να εξασφαλίσετε αυτό που υποτίθεται ότι είναι προστασία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Κομισιόν. Πρέπει να εξηγήσουμε πολύ περισσότερα και τα συμφέροντα των τοματοπαραγωγών μας πρέπει να προστατευθούν. Αλλά να πω και το εξής που πρέπει να είναι σαφές. Έχουμε αρκετές πολιτικές ανασφάλειες στη Βόρεια Αφρική. Το Μαρόκο είναι μια σταθερή χώρα στην περιοχή. Εάν δεν δώσουμε δυνατότητα στους Μαροκινούς να έχουν καλές εμπορικές σχέσεις μαζί μας και να τις αναπτύξουν, ούτω ώστε να βελτιωθεί η οικονομία του Μαρόκου εάν δεν εισαγάγουμε τα προϊόντα τους, τότε θα έρθουν αντί για τις ντομάτες οι νέοι από το Μαρόκο. Πρέπει λοιπόν να τους επιτρέψουμε να παράγουν προϊόντα που να μπορούν να μας τα πουλήσουν γιατί αλλιώ θα έρθουν οι ίδιοι. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε καλές συμφωνίες με τους Μαροκινούς. Και νομίζω ότι η Κομισιόν κάνει ό,τι μπορεί ούτως ώστε να προστατεύσει, να λάβει υπόψη και τα συμφέροντα των δικών μας παραγωγών. Δεν βλέπω να θέλει άλλο κάνει το λόγο. Οπότε ξαναδίνω το λόγο στην ε, Διευθύντρια. Ευχαριστώ. Όντω όπω είπατε, η συμφωνία είναι συμφωνία για, γεωργικές, για γεωγραφικές συγγνώμη, ενδείξεις προς, και την προστασία τους. Οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι όλα τα σήματα που σχετίζονται με προέλευση, ελεγχόμενη προέλευση, ε, ονομασία προελε... προστατευμένη ονομασία προελεύσεως κτλ. Αποτελούν ένα είδος ε, προστασίας της, ε, ενός δικαιώματος πνευματικής ιδιο... ιδιοκτησίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Επίτροπος μίλησε αυτή την εβδομάδα για ε, δικαίωμα αγροτικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. Δηλαδή συνδέεται ένα προϊόν με μια περιφέρεια. Η συμφωνία για παράδειγμα επιτρέπει κάθε γεωγραφική ένδειξη κρασιών, τυριών, άλλων γεωργικών προϊόντων όλα σχεδόν, όλες σχεδόν οι γεωργικές ενδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προστατεύονται στο Μαρόκο. Δεν μπορεί δηλαδή να καλέ, να αποκαλέσει ένας ε, παραγωγός του Μαρόκου το κρασί του Ριόχα, που είναι προστατευμένη. Αυτό είναι ο στόχος της συμφωνίας. Τώρα, για τις ντομάτες. Το πρόβλημα είναι ένα άλλο. Το πρόβλημα της ντομάτας είναι άσχετο με τη συμφωνία. Οι συζητήσεις που είχαμε για τον καθορισμό του υπολογισμού της αξίας στο τελωνίο της ντομάτας συνδέονται με αλλαγή της βασικής νομοθεσίας ε, μετά από τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής, μεταρρύθμιση η οποία εισήγαγε έναν υπολογισμό βάση καταποκοπή τιμής εισαγωγής. Με βάση αυτή την τιμή καταποκοπή διορθώθηκε η μέθοδος υπολογισμού της τιμής της ντομάτας κατά τη στιγμή της εισόδου στην αγορά της Ένωσης και συμπεριλήφθηκε στην τιμή αυτή όπως το απαιτεί ο κανονισμός, ένας υπολογισμός διαφόρων τύπων ντομάτας που μπαίνουν. Όχι οι κανονικές στρογγυλές ντομάτες, αλλά και τα, οι ντομάτες τσέρι, που είναι λίγο, οι μικρές ντομάτες δηλαδή, που είναι λίγο πιο ακριβές. Αν η τιμή παραγωγή είναι ψηλότερη της ε, τιμής εισόδου, δεν επιβάλλεται ε, δασμός. Αν η τιμή είναι χαμηλότερη από τη τιμή εισόδου, υπάρχει ένα δασμό, ένα ποσό δασμού. Αυτή τη στιγμή η τιμή εισόδου είναι 46,1 ευρώ τα 100 κιλό. κιλά. Αυτή είναι η τιμή εισόδου για το Μαρόκο. Η καταποκοπή τιμή εισαγωγή υπολογίζεται κάθε μέρα και όπως σας είπα είναι συγκρίσιμη. συγκρίνεται με την τιμή εισόδου. Αν είναι χαμηλότερη επιβάλλεται δασμό, αν είναι ανώτερη δεν εφαρμόζεται δασμό. Αυτά. Αλλά είναι άλλο θέμα αυτό. Δεν σχετίζεται δηλαδή με το ζήτημα των γεωγραφικών ενδείξεων και της σχετική συμφωνίας που σας παρουσίασα εδώ. Είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε κυρία Βουλευτής να σας δώσω περισσότερες εξηγήσει σε άλλο πλαίσιο. Σας ευχαριστούμε κυρία Διευθύντρια. Ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό. Ευχαριστούμε και για την παρουσία σας και για την ενημέρωση. Περνάμε στο επόμενο θέμα που αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Πρόκειται για ένα σημαντικό σχέδιο της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πολύ γρήγορα υποβλήθηκε. Ε, παρουσιάστηκε από τον Ιανουάριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στόχο έχει να αναζωογονήσει το επενδυτικό πρόγραμμα ήδη από τις 13 Ιανουαρίου υποβλήθηκε και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Αρμόδιες επιτροπές για το θέμα αυτό είναι οι επιτροπές ε, οικονομικών υποθέσεων και προϋπολογισμών και με αυτές θα συνεργαστούν βάσει τον άρθρο 55 ενώ οι επιτροπές βιομηχανίας και μεταφορών θα συνδεθούν με τις υπόλοιπες με βάση το άρθρο 54. Έχουμε και τον κανόνα 53 συν προκειμένου να υποβληθούν γνωμοδοτήσεις και από άλλες επιτροπές. Εμείς ε, ορίσαμε εισηγητή τον κύριο Αλμπερντές που θα συντάξει τη γνωμοδότησή μας για αυτό το πολύ σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα το γνωστό επενδυτικό πακέτο του κυρίου Γιούγκερ, του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ζητήσαμε να συμπεριληφθούν στο σημαντικό αυτό πακέτο και η γεωργία και η μεταποίηση, κάτι που παραλυπόταν στην αρχή. Κύριε Εισηγητά, κύριε Ντές, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που ως Επιτροπή Γεωργίας μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε. Η έκθεσή μου χαιρετίζει το ότι το σχέδιο Juncker προτείνει να γίνουν επενδύσεις στη γεωργία, στην Ήπεθρο και σε διάφορους σχετικούς τομείς. Η κοινή γεωργική πολιτική είναι ο καλύτερος τρόπος ούτως ώστε το Ταμείο αυτό να προωθήσει προγράμματα για την Ήπεθρο. Σημαντικό είναι το πρόγραμμα αυτό να εφαρμοστεί με μη γραφειοκρατικό τρόπο Έχω την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Το πρόγραμμα Juncker μπορεί να συμβάλλει για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, θέσεις εργασίας στην Ήπεθρο, συμπληρωματικές. Πρέπει να απαιτήσουμε η έρευνα και η καινοτομία να βοηθήσουν στην πρόθεση μιας βιώσιμης γεωργίας η έκθεσή μου θα περιέχει επίσης αναφορές για τις μειονεκτικές περιοχές και τις ιδιαίτερα περιφερειακές περιοχές και για την ανάγκη έκτακτης χρηματοδότησής τους. Στην έκθεσή μου θα προτείνω μέχρι 10 σημεία και θα σας την υποβάλω τις επόμενες μέρες γραπτός και θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να εκφράσουν τις επιθυμίες τους αλλά δεν πρόκειται να γράψουμε τώρα μυθιστόρημα θα αναφέρουμε μερικά σημεία Τώρα, επί της διαδικασίας. Η συζήτηση θα πρέπει να γίνει στις 24 Μαρτίου, προθεσμία για τροπολογίες. Μου υπόθηκε ότι είναι 25-26 Μαρτίου, αλλά θα έχετε πριν τη συζήτηση ήδη την έκθεσή μου γραπτός για να υποβάλλετε τροπολογίες. Ψηφοφορία στην Άγκρη 26 Απριλίου, στους προπολογισμούς 30 Απριλίου και έτσι έχουμε ένα καλό χρονοδιάγραμμα και ελπίζω η γνωμοδότηση αυτή να συμβάλλει το, σχέδιο Juncker να λάβει υπόψη τα συμφέροντα της Γεωργίας και της Υπέθρου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρθη ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ κύριε Κάρθη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ με τον εισηγητή. Είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή μας να προβάλλει μια πολύ στεναρή γνωμοδότηση. Ρωμαλαία. 315 δις σχέδιο επενδύσεων. Θα ενθουσιαστείς. Αλλά από τότε που αναγγέλθηκαν έχουν υποβληθεί πολύ περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις για το τι εννοεί η Επιτροπή. Πώς θα υπάρξει μόχλευση από τον ιδιωτικό τομέα. Και όλοι οι ευρωβουλευτές σίγουρα θα έχουν αρχίσει να λαμβάνουν email από πανεπιστήμια, άλλους φορείς, γιατί χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Κομισιόν. Αλλά υπάρχουν ε, μερικά στοιχεία που πρέπει να προωθήσουμε. Πρέπει οπωσδήποτε η Γεωργία να μην αδικηθεί. Σημαντικό είναι όμως επίσης, όπως είπε και ο συγητής, οι κοινότητες στην Ήπεθρο και αυτές που είναι ιδιαίτερα απομακρυσμένες να μην αδικηθούν. Άκουσα τον επικεφαλής της ΕΤΕ στην ΕΚΟΝ ότι στοχεύουν να υπάρχει η καλύτερη χρήση των πόρων. Αλλά κάποιες αποφάσεις πρέπει να έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Αν θέλουμε να επιτύχουμε πραγματικά τους στόχους μας, πρέπει όχι απλά να ευνοήσουμε μέσω των χρηματοδοτήσεων τις χώρες που επλήγησαν από την κρίση, αλλά κυρίως τις πιο μειονεκτικές περιοχές και περιφέρειες αυτών των χωρών. Εκεί που πραγματικά δεν υπάρχουν επενδύσεις, απασχόληση κτλ. Αυτό πρέπει να προωθήσουμε. Αυτά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αν είστε και μέλος της Επιτροπής ΕΚΟΝ, τότε γνωρίζετε πολύ καλύτερα πώς λειτουργεί αυτό το ταμείο και πώς θα δημιουργήσει μόχλευση, πώς θα προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια. Είστε πολύ καλύτερα κατατοπισμένος. Και αναφέρθηκε και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αλλά αυτό δεν είναι της δικής μας επιτροπής. Ο κύριος Σαν. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αφήνω το, τους αρμοδίους να δώσουν τις απαντήσεις και να αποφασίσουν ε, από πού θα προέρθουν αυτά τα χρήματα και με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτήσουμε αυτό το επενδυτικό πακέτο. Εγώ θα επικεντρωθώ σε άλλα θέματα, μια και είμαι ε, νέα εκλεγής ε, σκιώδης εισηγητής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για το θέμα αυτό. Και θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον κύριο Ντες ότι και η ομάδα μας ενδιαφέρεται για τα ίδια θέματα και μια και υπάρχει πίεση χρόνου προσβλέπω σε αγαστή και στενή συνεργασία και σας διαβεβαιώ ότι είμαι απόλυτα πρόθυμος γι' αυτό. Η ομάδα μου, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες, είναι αποφασισμένοι να σας βοηθήσει για να διαμορφώσουμε πραγματικά ηχηρά πολιτικά μηνύματα και ρωμαλαία. Εγώ θα σταθώ σε δύο ζητήματα. Το θέμα αφορά την προσθετικότητα, τη συμπληρωματικότητα. Πρόκειται για νέα ε, για, για κονδύλια που θα πρέπει να πραγματικά να έχουν προστιθέμενη αξία ε, και να ενισχύσουν, να αναβαθμίσουν τα ισχύοντα προγράμματα. Και πέραν ε, των κλασικών τομέων που τόνισε ο κύριος Δες, θα πρέπει να εξάρουμε και τη σημασία της αγροτικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης της υπαίθρου, επίσης της ενεργειακής απόδοσης, της ισορροπίας μεταξύ των κρατικών επενδύσεων και των ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτά τα θέματα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους σοσιαλιστές. Και εγώ, ως πραγματικός φίλος της εκπαίδευσης, ε, της έρευνας ε, και της γνώσης ε, που θα πρέπει να φτάσουν μέχρι την Ήπεθρο. Θα φροντίσω να ληφθούν όλα αυτά υπόψη. Και επίσης χρειαζόμαστε και διαφάνεια και τις ευρυζωνικότητα που θα πρέπει να φτάσει μέχρι την Ήπεθρο. Χρειαζόμαστε λοιπόν διαφάνεια για το πώς θα βρεθούν αυτά τα κονδύλια και πού θα διοχετευτούν. Γιατί αυτό το θέμα ενδιαφέρει ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης το θέμα της πάταξης της διαφθοράς. Οι περισσότερες φορολογικές απάτες και φοροδιαφυγές σχετίζονται με το τομέα των τροφίμων. Αυτά είναι θέματα που μας ενδιαφέρουν και προστίθενται σε όσα μας ανέφερε ο κύριος Δες. Και μαζί και με τους άλλους συναδέλφους από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα συνεργαστούμε για να επισπεύσουμε την διαδικασία και να καταλήξουμε σε μια πολύ μεστή γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σφεράου. Ναι, ευχαριστώ. Όλοι γνωρίζετε ότι ο κ. Γιούνκερ είναι ειδικό τη επενδύσει. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Τι κρύβεται πίσω από αυτό το σχέδιο στρατηγικών επιδιώσεων των 350 δις ευρώ. Νομίζω ότι το σχέδιο Juncker δεν, δεν, ε, δεν δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για τη γεωργία. Ε, πολύ μικρό κομμάτι των στρατηγικών επενδύσεων καλύπτεται από αυτό. Το θέμα της ε, πολεμικής αυτής είναι ξεκάθαρο. Γιατί δεν προωθήθηκε περισσότερο η γεωργία όπως οι υποδομές, οι νέες τεχνολογίες. Έχει τρομερές δυνατότητες. Φερρυπίν, την προστιθέμενη αξία και την, τις ονομασίες προελεύσεως, το δυναμικό των οποίων υπό, την χάνει υπό εκμετάλλευση στην Ευρώπη σήμερα. Γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε αυτό που έγινε με το κρασί, που για πολλές χώρες όπως η Γαλλία αποτελεί ένα μεγάλο ατού στην παραγωγή. Στο σχέδιο Γιούνκερ υπάρχουν πολλά να πούμε. Αυτό που θα πρέπει ωστόσο να τονίσουμε είναι ότι η γεωργία δεν βρίσκεται στο ύψος των απαιτήσεων για τέτοιες επενδύσεις. Και εγώ παρόμοια ερώτηση είχα υποβάλει και η απάντησή μου ήταν ότι η κοινή γεωργική πολιτική είναι εφοδιασμένη με πολλά κονδύλια. και σίγουρα ε, μου είπαν ότι αγαπούν τη γεωργία, αλλά δεν είναι ο μόνος οικονομικός κλάδος, υπάρχουν και άλλοι οικονομικοί τομείς. Ο κύριος Ροπέ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το σχέδιο αυτό το έχουμε συζητήσει πολύ. Τώρα είναι ηρεμότερο το κλίμα και γι' αυτό είμαι αισιόδοξο. Ελπίζω λοιπόν το σχέδιο Γιούγκερ να επιτύχει Ελπίζω να μεταγραφεί σε συγκεκριμένα μέτρα και η στόχη μας είναι η οικονομική ανάπτυξη και θέσει απασχόλησης. Είναι αναγκαία η απασχόληση. Και η γεωργία είναι τομέας όπου χρειαζόμαστε απασχόληση. Έχει πολλές δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας σε πολλά κράτη-μέλη, για παράδειγμα, μπορούμε να επιτύχουμε πολλά δημιουργώντας ε, θέσεις εργασίας στο βόηο τομέα και σε άλλους τομείς. Για να αυξηθεί και ο πληθυσμός. Και ε, αν αυξηθεί ο πληθυσμός θα χρειαστούμε περισσότερο, περισσότερα τρόφιμα και βεβαίω πρέπει να ε, αυξήσουμε και τι δυνατότητες εξαγωγής ποιοτικών τροφίμων. Πρέπει να αποκτήσουμε πρόσβαση σε νέες αγορές. Αυτό επίσης θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Επίση, θεωρώ ότι το σχέδιο αυτό θα έπρεπε οπωσδήποτε να ασχοληθεί και με τις υποδομές της υπαίθρου. Για παράδειγμα, τις ανακαινήσεις ε, κατοικιών. Ήδη γίνεται. Όμως δεν γίνεται παρκώς στην Ήπεθρο. Εδώ πρέπει να έχουμε ανακαίνιση ε, των κατοικιών. Διότι αυτό θα βοηθήσει την παραμονή του πληθυσμού στην Ήπεθρο, αν έχουν καλύτερη κατοικία. Και θα δημιουργήσει και θέσεις εργασίας ακριβώς εκεί μέσω της ανακαίνησης. Επίσης ε, η πράσινη ενέργεια το βιοαέριο. Όλα αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτό το νέο πλαίσιο. Θα το καλωσορίσουν και οι γεωργοί και θα δώσει δυνατότητες και επενδύσεων για το ιδιωτικό κεφάλαιο. Και βεβαίως ε, πρέπει στη συζήτηση να συμπεριληφθούν και οι περιφέρειες για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν λόγο. Η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Η επιτυχία του, των στρατηγικών επενδύσεων εξαρτάται από το αν τα κράτη-μέλη υποβάλλουν project. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του κ. Δες ε, σε κάποιε από τι λεπτομέρειε τη πρότασή του. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πού βρίσκονται. Πρέπει να υπάρχουν επενδύσει στην ευρυζωνική ε, στο ευρυζωνικό φάσμα, ε, αντικαθιστώντας τι εθνικέ επενδύσεις. Βέβαια, δεν ξέρω αν η εντολή αυτή μπορεί να καλύψει τα πάντα, γιατί τα project υποβάλλονται, όπως σας είπα, από τα κράτη-μέλη. Εμείς πώς κολλάμε. Το πρόγραμμα αυτό δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να αντικαταστήσουμε την κοινή γεωργική πολιτική. Πρέπει να υπάρχουν και άρα χρειάζεται ε, προσθετικότητα. Το ξέρουμε αυτό. Πριν δούμε κάποιες ιδέες στην έκθεση, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κρίνουμε αν μπορούμε να συμβάλλουμε στη συζήτηση ως Επιτροπή Γεωργίας. Προφανώς ωστόσο υπάρχουν τομείς όπου οι κοινότητες υπαίθρου χρειάζονται επενδύσεις. Το επιχείρημα ωστόσο είναι ότι οι αυτοκινητόδρομοι και τέτοιες επενδύσεις βοηθούν όλους και τις περιφέρειες. Τα καλά έργα είναι αυτά που χρειάζονται. Ευχαριστώ. Ε, φυσικά τα κρατη μελη θα αποφασίσουν ε, ποια σχέδια θα επιλέξουν. Ο κύριος Νταντά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε μεμονωμένες επενδύσεις στην Ήπεθρο. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε οι επενδύσεις αυτές ε, να στηρίξουν ένα ολόκληρο κλάδο είτε τη γεωργία είτε τη δασοκομεία. Δεν μπορούμε να λέμε ότι το σχέδιο Juncker, το επενδυτικό, θα πρέπει να συμβάλλει ε, ε, στην βελτίωση ενεργειακής απόδοσης αν δεν στηρίξουμε ολόκληρο κλάδο. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη σε ό,τι αφορά την στήριξη των επενδύσεων της υπαίθρου. Τώρα, στην Ήπεθρο, συγγνώμη, για, τη, για τον ψηφιακό αλφαβητισμό. Σίγουρα οι χώρε που επενδύουν στην ευρυζωνικότητα, για παράδειγμα στην Ήπεθρο, ξεκινούν από τι πιο πυκνοκατοικημένε ε, περιοχέ τη Ήπεθρου. Και μάλιστα έχουμε κάποιες ορεινές περιοχές που αν ε, δεν εξασφαλίσουμε πρόσβασή τους στον ψηφιακό κόσμο θα είναι τελείως αποκομμένες ε, γιατί καμία επιχείρηση δεν θα θέλει να προσφέρει υπηρεσίες εκεί. Μόνο κινητοποιώντας μέσα και στηρίζοντας οικονομικές πρωτοβουλίες μπορούμε να αποφύγουμε κατακαιρματισμό των ευρωπαϊκών περιφερειών και διαχωρισμό μεταξύ εκείνων που έχουν πρόσβαση στα πάντα και εκείνων που δεν έχουν πρόσβαση σε τίποτα. Παρακαλώ κύριος Ντες. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για τις παρεμβάσεις σας. Βεβαίως σημείωσα επιμελώς να συνοψίσω για τον πρώτο ομιλητή. Βεβαίως ακόμη συζητείται η χρηματοδότηση, αλλά δεν είναι αυτό το καθήκον μου. Εφόσον έχουμε το πρόγραμμα Juncker, εμάς μας ενδιαφέρει να αξιοποιηθεί και προς το συμφέρον ε, της γεωργίας και της Υπέθρου και νομίζω ότι θα επιτύχει. Φυσικά θα τα ξανασυζητήσω με τους σκιώδεις, δεν το είπα προηγουμένως, είναι αυτονόητο. Οπωσδήποτε και την έκθεση και το ψήφισμα θα τα συμφωνήσω μαζί τους. Να τονίσω ιδιαίτερος <clears throat> ότι οι επενδύσεις σε υποδομές είναι αποφασιστικές. Το είπαν οι Μαγκίνες και ο Νταντά. Για παράδειγμα, ευρυζωνικότητα. Πολύ σημαντικό. Μπορούμε να αναφέρουμε συγκεκριμένα σημεία αλλά δεν θέλω τώρα να κάνω ολόκληρο αναλυτικό κατάλογο. Πρέπει να περιοριστούμε στα κυριότερα αιτήματα. Και τα κυριότερα αιτήματα είναι οι επενδύσεις να γίνουν στις οικονομικά αδύναμες περιοχές. Στην περιοχή μου έχουμε 2% ανεργία. 0% ανεργία των νέων. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν επενδύσεις εμείς. Οι επενδύσεις πρέπει να γίνουν εκεί που υπάρχει υψηλή ανεργία των νέων στην Ήπεθρο εκεί που υπάρχει υψηλή ανεργία γενικότερα. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτές οι περιφέρειες πρέπει να επανασυνδεθούν με την οικονομική ανάπτυξη. Η περιφέρειά μου μετά τον πόλεμο ήταν ιδιαίτερα μειονεκτική. Μέσω εγκαίρων επενδύσεων σε υποδομές, μπορώ να το επιβεβαιώσω, η περιοχή μου είναι πρωτοπόρα σήμερα στη Βαβαρία. Λοιπόν, διότι οι πολιτικοί πριν από 40-50 χρόνια έλαβαν τις σωστές αποφάσεις. Θα ήθελα λοιπόν να γίνει αυτό και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, ούτω ώστε να υπάρξει επαρκής οικονομική ανάπτυξη και από πλευράς ε, της δικής μας αρμοδιότητας θέλουμε οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί η Ήπεθρος. Ευχαριστώ τον ε, Πρόεδρο Σικέρσκι γιατί έπαιξε ρόλο στις προκαταρκτικές ε, επαφές που κάναμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό και στην επόμενη συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου. Θα το ξανασυζητήσουμε και στο μεταξύ αν έχετε συστάσεις ή προτάσεις ε, αποταθείτε στον κύριο Ντές ε, για να τις υποβάλλετε. Θα συνεχίσουμε, επαναλαμβάνω, τη συζήτησή μας ε, στις 23 Μαρτίου, στην επόμενη συνεδρίαση. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο, τις συστάσεις των συντονιστών. Έχετε λάβει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τις ε, προτάσεις των συντονιστών, αλλά και έγγραφο. Είναι η αποφάση της πρωινής συνεδρίασης οι συστάση μάλλον της πρωινής συνεδρίασης και αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις ε, θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένες. Δεν βλέπω αντιρρήσεις ε, για τις συστάσεις των συντοριστών, οπότε εγκρίνονται και περνάμε στα διάφορα. Δεν υπάρχουν διάφορα. Επόμενη συνεδρίασή μας στις 23 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα, 3 το απόγευμα και 24 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη, πρωί και απόγευμα. Αυτά διεκπαιρεώσαμε την ημερήσια διάταξη. Μερικά θέματα τα αφήσαμε για την επόμενη συνεδρίαση. Ευχαριστώ και ραντεβού στην επόμενη συνεδρίαση σε ένα περίπου μήνα. Στο μεταξύ έχουμε άλλα, άλλες δουλειές ο καθένας. Ευχαριστώ. Λύεται η συνεδρίαση.